Να ξεκινήσουμε. Καλώ ήρθατε όλοι. Πάνω απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνεδρίασή μα τη Επιτροπή, Ευχόμενος χρόνια πολλά στον κύριο Κόστιγκερ. Χρόνια πολλά. Στην κυρία Κόστιγκερ. Και μετά ήθελα να χαιρετήσω επίση τους παραγωγούς γάλακτος της περιοχής spider Α, δεν έφτασαν ακόμα. Όταν, ε, όταν έρθουν κάντε μου ένα σήμερα. Ούτω ώστε να χαιρετήσω. Τι παράγουν γάλα και γκράπα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας με το πρώτο σημείο την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν κάποιε παρατηρήσεις θεωρούμε την ημερήσια διάταξη εγκεκριμένη. Έχω τη χαρά να σας πω ότι η διερμηνία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της Επιτροπής μας. Ωραία. Μετά σημείο 2, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 26ης Σεπτεμβρίου, 5 και 6 Οκτωβρίου και 12 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θέλω συνεδριάσεως και τα πρακτικά τα θεωρούμε ως συγκεκριμένα. Η σημερινή συνεδρίαση μεταβιβάζεται και μέσω διαδικτύου με το web stream. Θα ήθελα να επιθυμήσω ότι αύριο το απόγευμα η Πολωνική Προεδρία σε συνεργασία με την Επιτροπή μας, πρωτοβουλία όμως είναι της Πολωνικής Προεδρίας, θα διοργανώσει μια ακρόαση με τις επαγγελματικές οργανώσεις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αίθουσα Τζαν 2Q2 Υπάρχουν πολλές ε, οργανώσεις που προσεκλήθησαν από την Πολωνική Προεδρία. Εμείς ε, βοηθάμε, αλλά είναι μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Υπουργό Μάρεκ Ζαβίνσκι και από την Πολωνική Προεδρία. Βλέποντας πώς οι οργανισμοί προσεκλήθησαν, μόνο οι συγητές πιθανότατα θα μπορούσαν να πάρουν το λόγο. Μετά όμως θα δούμε κατά τη των εργασιών, αν θα υπάρξει δυνατότητα ενδεχομένως να πάρουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι που θα θελήσουν να μιλήσουν σας ανακοινώνω ότι είναι μια πρωτοβουλία που ήθελε να διοργανώσει η Πολωνική Προεδρία με τη βοήθειά μας και υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις, γεωργικές συνεταιρισμοί, ε, νέοι γεωργοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πάρα πολύ προσκεκλημένη θα είναι. Αυτό θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα. Λοιπόν, δεν έφτασαν ακόμα η γαλακτοπαραγωγή της περιοχής πάει. Όχι. Πάμε στο σημείο 4. Είναι ένα σημαντικό σημείο τη ημερήσια διάταξη. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ορισμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση αξιολόγηση του αντικτύπου τη κοινή αγροτική πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει σε εμά κάποια θέματα τη αξιολόγηση αντικτύπου και βεβαίως θα απαντήσει στα σχόλια και στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Τα θέματα που καλύπτονται και θα άτομα τη ευκαιρία χαιρετήσω τον κύριο Τάσο Χανιώτη που είναι ο διευθυντή και είναι μαζί μας, μαζί με άλλους φίλους που δεν ξέρω αν του βλέπω όλου, αλλά είναι και άλλοι, ναι, σας χαιρετώ. Τα σημεία είναι greenings, πράσινη χρειά, η ανακατανομή των πληρωμών της ΚΑΠ, εδεχομένη τομής δικαιώματο ε, ενίσχυση σταδιακή μείωση των άμεσων πληρωμών και τέταρτο σημείο, το ΚΙΤ, τα εργαλεία της διαχείρισης του κινδύνου. Επ' αυτών των τεσσάρων ε, σημείων, ο Τάσος Χανιώτης και άλλοι φίλοι της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας θα, θα αναφερθούν σε αξιολόγηση του δικτύπου και θα ακούσουμε αμέσω τι έχουν να μας πούν και θα σημειώσουμε και επίση ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Τάσο, 20 λεπτά για την παρουσίαση και θέλω να αφήσω περιθώριο χρόνο γιατί σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις των συναδέλφων. Έχει το λόγο η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας λοιπόν. Ορίστε. Thank you, Chairman. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη. Τάσο, θέλω να τους χαιρετήσω όλους τους γαλακτοπαραγωγούς της περιοχής. Είναι πάνω από 40 γαλακτοπαραγωγοί της ΠαΐΕΡΒΕ που ε, θέλω να τι χαιρετήσουμε και του ευχαριστήσουμε για την παρουσία του μαζί και με τον κύριο Μάρκ Ταραμπέλα που του κάλεσε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και καλώ ήρθατε. Λοιπόν, έχει το λόγο, Τάσο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, για να κερδίσουμε χρόνο, θα είμαι σύντομος. Αυτό που σας παρουσιάσω σήμερα είναι μια σύνοψη δύο παρουσιάσεων που κάναμε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου. Η μία που έχει να κάνει με θέμα που αφορά στη διανομή, κατανομή των πόρων και το άλλο ε, έχει να κάνει με τη γενική ε, εικόνα και προοπτική της αγοράς. Θα αρχίσω από αυτό το δεύτερο γιατί υπάρχουν ε, ορισμένα νέα στοιχεία που εντάσσονται ε, στην πρόβλεψη των αργορών μέχρι το 2020. Θα σας δώσω μερικές παραδοχές ε, που χρησιμοποιήσαμε στη σύνοψη και βεβαίως θα επηρεάσουν ε, και τη συζήτηση για ορισμένα από τα μέτρα που προτείνουμε. Και το δεύτερο, ιδιαίτερα θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη αντικτύπου και ιδιαίτερα αυτά που έχετε τονίσει κι εσείς. Θα ήθελα να διευκρινίσω από την αρχή ότι στη μελέτη αντικτύπου δεν μελετήσαμε αποκλειστικά ε, τις ε, εναλλακτικές προτάσεις. Γενικά κάναμε κάποιες παραδοχές και κάποιες ε, αντιστοιχίες, αλλά όχι ένα προς ένα. Αρχίζω από τις προοπτικές της αγοράς. Φέτος είχαμε μια διαφορά σε σχέση με τα όσα είχαμε στο παρελθόν. Ήδη από πέρσι αρχίσαμε την μεσοπρόθεσμη εξέταση. Ε, το καλοκαίρι ε, είχαμε τα στοιχεία της εσοδείας από το Βόρειο Εμισφαίριο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, προσθέσαμε και τη βραχυπρόθεσμη εκτίμηση για τις γεωργικές αγορές. Αυτό σας το είχε υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του G20 για να αυξηθεί η διαφάνεια και η λειτουργία των παγκόσμιων αγορών και το ακολουθήσαμε και εμείς. Και τέλος, Χρησιμοποιήσαμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία από συναδέλφους της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΦΙΝ οικονομικών αλλά και από άλλες πηγές ε, ε, με πιο μακροπρόθεσμα στοιχεία. Uh, Για να σας πω πώς έχει η οικονομική κατάσταση. Εδώ το μπλε στη γραφική παράσταση είναι η αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαρτίου 2008 πριν ξεσπάσει μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση. Και το πορτοκαλί είναι η πραγματική τελικά κατάσταση και βλέπετε ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στα εκτιμόμενα αποτελέσματα και στα πραγματικά και τις προβλέψεις. Αυτή η διαφορά στις προβλέψεις προφανώς έχει επιπτώσεις και στη ζήτηση γεωργικών προϊόντων αλλά και στην προσφορά. Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά που βλέπουμε εδώ σε αυτή την εικόνα ε, εμφανίζεται σε τούτη εδώ τη γραφική παράσταση που είναι η αλλαγή και η εξέλιξη των παγκοσμίων τιμών ε, γεωργικών ε, προϊόντων, ενέργειας και λοιπασμάτων είναι οι δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας και βασίζεται σε μια εκτίμηση. Βλέπετε μέχρι το 2004 από το 1996, από το 86 μάλιστα ήταν κάπως σταθερή εξέλιξη. Από το 2004 αυξήθηκαν πάνω από 60%, ε, τριπλασιάστηκαν ε, τα λοιπάσματα και τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με τα γεωρικά προϊόντα, οι τιμές της ενέργειας. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τι δείχνουν, ότι η κατάσταση για το ε, πώς θα ανταποκριθεί η γεωργία σε αυτές τις προκλήσεις είναι πιο περίπλοκη. Με τις σημερινές τιμές, οι τιμές υποστήριξης της αγοράς δεν παίζουν κανένα ρόλο ή μάλλον ευτερεύοντα, και αυτό που αποκτά μεγαλύτερη σημασία είναι το στοιχείο του κόστους και οι ανάγκες να προσαρμοστεί η γεωργία σε αυτές τις προκλήσεις. Μεγάλη διαφορά που βλέπουμε στη ζήτηση των ε, δημητριακών εμφανίζεται εδώ. Αν κοιτάξετε τις ε, ε, γραμμές και εισαγωγές και εξαγωγές περίπου αναμένονται να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα. Δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές ε, στις ζωοτροφές, στη ζήτηση ή για μη ε, χρήση ζωοτροφών, αλλά τα βιοκαύσιμα είναι εκείνα που έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσει για τα σιτήρα. Το είδαμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγα χρόνια και ακριβώς εκεί. Τώρα στις αρωτρές καλλιέργειες ε, είπαμε τα βιοκαύσιμα και πραγματικά οι τιμές ε, αναμένονται ψηλές. Οι εσοδίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται με χαμηλότερο βαθμό ε, από ό,τι στις άλλες ανταγωνίστριες ε, περιοχές. Ε, ο αραβόσιτος και το μαλακό σιτάρι θα συνεχίσουν να καλύπτουν το έδαφος και οι ελαιούχοι σπόροι αυξάνονται με χαμηλότερο αριθμό και βλέπουν και κάποια αύξηση στην παραγωγη ζάχαροτεύτλων. Αυτό έχει να κάνει το γεγονός ότι στη Βραζιλία πολύ ζάχαρη πηγαίνει για καύσιμα ε, στα αυτοκίνητα, οπότε έχουμε κάποιο χώρο εκεί για τα ζαχαρότευτα στα κρέατα τώρα. Ε, αυξάνονται οι ανάγκες και η ζήτηση, γι' αυτό σε μια κατάσταση ε, που παραμένει σταθερή η ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα είμαστε ε, στο μέλλον καθαρή εξαγωγής πουλερικών και χειρίου κρέατος. Έτσι έχουμε δει τις εκτιμήσεις αυτές στην αγορά πουλερικών. Επίσης ε, για το γάλα υπάρχει κάποια ε, μεγαλύτερη ζήτηση και μικρή αύξηση στην προσφορά και υπάρχει δυνατότητα εξαγωγών γαλακτοκομικών ε, προϊόντων, αλλά το μερίδιό μας στην αγορά παραμένει χαμηλό γιατί άλλοι αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς. Αυτά ήταν πραγματικά με δύο λόγια ως προς την κατάσταση της αγοράς. Τι κάνουμε τώρα με τη μελέτη σκοπιμότητας. 20 γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν σε μια προσπάθεια σε μια άσκηση που άρχισε τον Απρίλιο του 10 και τελείωσε τον Ιούνιο του 2011 είχαμε εκτενέστατες διαβουλεύσεις πάνω από 517 απαντήσεις του κοινού και ήταν γενική η συνένεση ότι θα πρέπει να βασίζεται η κοινή γεωργική πολιτική στη δομή των δύο πυλώνων και με καλύτερη στόχευση περισσότερο πρασίνισμα εντό εισαγωγικών και μεγαλύτερη ολοκλήρωση και σωμάτωση τη κοινή γεωργική πολιτική μαζί με άλλε πολιτικέ. Μεθοδολογία τώρα. Εσωτερική ανάλυση και μικροοικονομική και πιο τομεακή. Είχαμε ένα διεθνές εργαστήριο που αξιολόγησε τα αποτελέσματα και τα σχολίασε και σε εμπειρογνώμονε από το USDA, οικονομολόγους ε, ή του ΦΑΟ, ε, του ΑΕΚ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και γενικά υψηλού επίπεδου. Είχαμε και από τις διαχειριστικές επιτροπές στοιχεία και οικονομικές και άλλες μελέτες Επίσης χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ εξωτερικές μελέτες και αναλύσεις για την κοινή γεωργική πολιτική. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τους στόχους ε, ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, ε, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτά και αποτελεσματικότητα ε, ήταν οι στόχοι της μεταρρύθμισης. Τρία γενικότερα σενάρια. Το σενάριο της προσαρμογής βασίστηκε στην αναγνώριση ότι η βασική αποτυχία πολιτικής του σημερινού συστήματος ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται οι ενισχύσεις, οπότε εστιάσαμε περισσότερο σε μεγαλύτερη ισότητα στις άμεσες πληρωμές, προσθέσαμε στη δεύτερη επιλογή που ονομάζουμε ολοκλήρωση integration τα στοιχεία του πρασινίσματος ε, του πρώτου πυλώνα που είναι η βασική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπήρξε και μια άλλη λύση, μια άλλη πρόταση που στην αρχή της συζήτησης γνώρισε μεγάλη προσοχή που ε, με υψηλές γεωργικές τιμές και αυτή την προοπτική θεωρήσαμε ότι δεν χρειάζεται ενίσχυση το εισόδημα των γεωργών, οπότε σταδιακά θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι άμεσες πληρωμές ένα μέρο των χρημάτων να επιστρέψει στου φορολογούμενους και το άλλο στο δεύτερο πυλώνα. Στην ανάπτυξη τη υπαίθρου. Αυξήθηκε όμως πολύ το κόστος των, ε, του input των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία πριν την παραγωγή, οπότε έχει εγκαταληφθεί μάλλον αυτό το σενάριο. Βλέπετε εδώ τη σύγκριση των διαφόρων σενάριων. Αναστόχο Γενικά, η επανεστίαση, το τελευταίο σενάριο, μαζί με αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στις πιο ανταγωνιστικές περιοχές θα σήμαινε ότι θα εγκαταλειφθεί η παραγωγή στις λιγότερο ανταγωνιστικές. Το άλλο σενάριο της ολοκλήρωσης της εσωμάτωσης δίνει αποτελέσματα γενικότερα πιο ισόρροπα, αλλά αυξάνεται κάπως και το διοικητικό κόστος. Σε ό,τι αφορά τώρα τα σενάρια αναδιανομής για τις άμεσες πληρωμές, εστιάσαμε σε δύο σημεία, αρχίζοντας από την αιτιολόγηση των αμέσων πληρωμών. Αυτό γίνονται για στήριξη του εισοδήματος, αλλά και για να έχουμε ένα βασικό δημόσιο αγαθό. Και προσπαθούσαμε να δούμε τι γίνεται με τη στραματική ενίσχυση με κριτήρια οικονομικά ή περιβαλλοντικά. Πώς διαμορφώνεται αυτό. Λοιπόν, ένα από αυτά τα σενάρια είναι αυτό που βλέπουμε στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Στις γαλάζιες στήλε βλέπετε πώς γίνεται ε, σήμερα η στραματική ενίσχυση ή ευρώ γινεται σημερα η στραματικη εκτάριο, εν περιπτώσει. Ε, το, η κόκκινη γραμμή είναι ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διάστηκτη ε, γραμμή διακεκομένη είναι που θα βρίσκονταν τα κράτη-μέλη εάν η κατανομή των ενισχύσεων ή ένα διανομή βασιζόταν στα 2 τρίτα του ΑΕΠ και στο 1 τρίτο στην προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα. Και ε, με κριτήρια περιβαλλοντικά, λίγο πιο περίπλοκος ο υπολογισμός, μας δίνει αυτή την εικόνα. Είναι κάπως διαφορετικό με τον προηγούμενο ε, ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η κατανομή των κονδυλίων. Αλλάζει. Θα βρείτε στα, παραδείγματα, στα παραρτήματα πολύ πιο λεπτομερείς πίνακες, με ποια κριτήρια δηλαδή καταλήξαμε σε αυτό τον υπολογισμό και τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται και κατατάσσονται ανακράτος μέλος. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από εδώ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να μην πω ανέφεκτο, να φτάσουμε σε μια αντικειμενική κατανομή των ενισχύσεων. Γι' αυτό προχωρήσαμε σε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση όπου βάσει του μέσου όρου ε, του κοινοτικού έχουμε βάλει ως στόχο την κάλυψη του ελλείμματος όρου μέχρι το 90% και τελικά το 1 τρίτο ε, καλύπτεται από τη βαρούσα πρόταση. Δεν είναι μυστικό ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει στη συζήτηση και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο πριν ληφθεί απόφαση, αλλά αυτή η πρόταση βασίζεται επίσης και στο γεγονός ότι δεν κοιτάμε μόνο τι γίνεται στον πρώτο πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής, αλλά έχουμε ένα πολύ ευρύτερο πρίσμα στη θεώρησή μας και στις θέσεις των κρατών μελών. Έρχομαι τώρα στο λεγόμενο πρασίνισμα της γεωργίας. μελετήσαμε πάρα πολύ το κόστος των διαφόρων αυτών μέτρων για το περιβάλλον και υποθέσαμε ότι σε κάθε υποπεριφέρεια, ε, στο δείγμα που είχαμε 18.000 εκμεταλλεύσεις, θεωρήσαμε ότι κάθε γεωργική εκμετάλλευση θα έπρεπε να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα για το περιβάλλον. Και υπολογίσαμε ότι το μερίδιο των ε, εκμεταλλεύσεων σε μέσο όρο στην Ένωση θα ήταν 80% ε, περίπου. Ε, με αυξημένο κόστος, κάποιο κόστος. Η Ιρλανδία είναι τόσο χαμηλά εκεί που βλέπετε γιατί έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μονίμων χορτολιβαδικών εκτάσεων, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα και το συνολικό κόστος της ε, πρασινίσματος σαν κράτος μέλος είναι σε αυτή τη διαφάνεια που σας δείχνω τώρα για την ε, κάλυψη σε πράσινο, σε λιβάδια, αλλά αυτό καταλήφθηκε ως ε, λύση γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Ο μέσος όρος της στραματικής ενίσχυσης ήταν 33 ευρώ ανά εκτάριο για κάθε επιλέξιμη ε, περιοχή και 41 ευρώ ανά εκτάριο μόνο για τις εκμεταλλεύσεις που πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλά είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές οι οποίες κρύβονται εδώ ε, και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα σε κλάδους παραγωγής που θα σας εξηγήσω αναλυτικά. Εδώ θέλω να φέρω το εξής, γιατί υπήρξε ήδη κάποια σύγχυση σε σχέση με ορισμένα από τα αποτελέσματα είναι και λογικό και φυσικό και αναμενόμενο γιατί είναι περίπλοκη η κατάσταση να δημιουργείται κάποια σύγχυση. Το κόστος, για παράδειγμα, μιας περιοχής με οικολογική εστίαση που έχουμε στα αποτελέσματα της ανάλυσης δίδεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το ένα είναι το κόστος ανά εκτάριο ή αναστρέμα που είναι πάνω από 260 ευρώ το εκτάριο και μετά το συνολικό που είναι μόλις 6 ευρώ ανά εκτάριο. Γιατί περίπου στη μισή επικράτεια δεν χρειάζεται να κάνει κανείς τίποτα και στην άλλη μισή ε, ε, χρειάζεται παρέμβαση. Έχουμε εδώ το χάρτη τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνει την αρχική κατανομή αυτού του κόστους. Όσο πιο πράσινο είναι το χρώμα, τόσο πιο υψηλό είναι το κόστος. Δηλαδή όταν είναι πιο σκούρο πράσινο, ξεπερνάει όπως βλέπετε τα 50 ευρώ ανά εκτάριο. Επίσης, κοιτάξαμε τι γίνεται και με τους μικρούς αγρότες, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, για να μην επηρεαστεί η δυνατότητα των μικρογεωργών να έχουν ένα πιο απλό σύστημα. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά σήμερα ε, στο μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη. Είναι εδώ οι πράσινες στήλες και ε, δεξιά βλέπετε το ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που είναι κάτω των 5 εκταρίων, ή 50 στρέμματα δηλαδή. Τώρα, σε αυτή εδώ τη διαφάνεια βλέπουμε τον προϋπολογισμό, πώς κατανέμεται και ποιος είναι ο αριθμός των μικρογεωργών που είναι οι τελικοί δικαιούχοι, εάν ε, είναι 50% το ποσοστό των κρατών μελών. Στο γαλάζιο βλέπετε πόσοι είναι οι δικαιούχοι κάτω από το κατόφλι. Ε, το, ε, το γαλάζιο χρώμα. Ενώ το μοβ δείχνει τα ποσά, τα πραγματικά ποσά, όχι τα ποσοστά. Μετά ε, τη Λετωνία, βλέπετε την Εστονία, όλα τα κράτη αριστερά της Λετωνίας είναι με χίλια ευρώ ανά μικρό γεωργό θα εξαντλούσαν τον προπολογισμό τους. Ενώ δεξιά από την Εστονία και πέρα δηλαδή, τα χρήματα στη διάθεσή τους ε, για να εκτελέσουν και να εξαντλήσουν τον προπολογισμό. Γι' αυτό ε, αυξήσαμε το κατόφλι αυτό στο 10% για να μπορούν τα κράτη-μέλη, εάν το επιθυμούν, να προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ για λόγους οικονομίας χρόνου. Με χαρά να απαντήσω σε οποιασδήποτε λεπτομερείς ερωτήσεις έχετε, είτε σήμερα είτε αργότερα. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Α, υπάρχει και ένα αναλυτικό παράρτημα ε, με περισσότερε διαφάνειε, το οποίο έχω αφήσει στην άκρη αλλά είναι στα χέρια σα να το μελετήσετε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ υλικό προσυζήτηση. συζήτηση. Έχουμε ήδη κατάλογο μεγάλο με παρεμβάσει. Θα ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Νικολέσκου και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλοι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Διευθυντά, για αυτή την παρουσίαση και θα έλεγα ότι η Επιτροπή μας δεν θέλει να μείνει εκτός παράμερα, ούτε το Κοινοβούλιο να μείνει εκτός. Έχουμε εκφράσει ήδη την άποψή μας σχετικά με το τι θέλαμε να δούμε σαν μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική. Το Κοινοβούλιο πάντα ζητούσε μεγαλύτερη η ισονομή στον αφορά τι αμέσω πληρονομέ στα κράτη-μέλη. Αυτό όμω δεν απορρέει από προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο αυτό που προτείνεται λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη Ρουμανία συγκεκριμένα δεν έχουμε υπόψη ότι αυτή η πρόταση θα πρέπει να υποστηριχθεί και θα ζητήσουμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε το 2015 λίγη ούτως ή άλλως η προθεσμία όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές και τις διαφορές. Πρέπει να είμαστε ισότιμοι με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και η Ρουμανία θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικ... μια σημαντική πηγή για την παραγωγή τροφίμων, πάντα βέβαια εφόσον ισότιμα θα αντιμετωπίζεται και δίκαια από τους εταίρους μας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δικαιολογείται αντικειμενικά λοιπόν αυτή η πρόταση, αυτά που προτείνονται και γι' αυτό αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας επεξηγήσει περισσότερο και καλύτερα πώς κατέληξαν σε αυτούς τους υπολογισμούς. Από πού άντλησαν αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Ρικουλέσκου. Πατράου Νεβές και μετά Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στο γεγονός ότι βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα μαζί μας περίπου 25 διευθυντές ε, της Συνομοσπονδίας ε, Παραγωγών Γεωργών της Πορτογαλίας. Δηλαδή, οι κυριότεροι εκπρόσωποι όλων των τομέων της παραγωγικής ε, γεωργίας της Πορτογαλίας. Και αυτό ακριβώς επειδή αφορά το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη που σήμερα βρίσκεται υπό εξέταση και διακυβεύεται. Και γιατί αυτό, διότι πιστεύουμε ειλικρινά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υλοποίησε μια θεμελιώδη υπόσχεση πρωταρχικού χαρακτήρα ευθύ εξ αρχή, δηλαδή για μεγαλύτερη ισότητα. Εμεί δεν βλέπουμε, εγώ δεν βλέπω μεγαλύτερη ισότητα σε αυτέ τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κατά τα άλλα επιτρέψτε μου να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στο γεγονό ότι ξεκινήσαμε να ε, κάνουμε λόγο, έγινε λόγος για την ανάγκη προσαρμογής της γεωργίας μας στις αγορές. Και ταυτόχρονα με υπογραμ... υπογραμμίζει το γεγονός ότι είναι χαμηλότερη η παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις υπόλοιπες περιφέρειες και περιοχές του κόσμου με τις οποίες ανταγωνιζόμαστε. Αυτές έχουν μεγαλύτερη αύξηση και ποσοστό αύξηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε ότι έχουμε περισσότερους κανόνες και κανονισμούς και επιβαρύνσεις να υλοποιήσουμε στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα δεν έχουμε μία ε, ας το πω έτσι, ιδιαίτερα ανθεκτική αγορά όσον αφορά τις εισαγωγές από άλλα μέρη του κόσμου. Με αυτό το σενάριο τώρα κάνουμε λόγο για μια ανακατανομή επιχορηγήσεων και υποστήριξης. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς με αυτόν τον τρόπο πώς η ισότητα θα μπορούσε ως αρχή να υλοποιηθεί με αυτές τις προτάσεις. Πράγματι αυτό που βλέπω είναι ότι όσον αφορά την Πορτογαλία διατηρούμαστε ακριβώς την ίδια κατάσταση που μέχρι σήμερα βρισκόμαστε. Δηλαδή στο 24ο ε, σημείο, στον 24ο βαθμό. Και όταν βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα είχε η Πορτογαλία τεράστιες διαφορές ε, και θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε 24η ε, σε 24η θέση, διαρωτώ με πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μάχη της ανταγωνιστικότητας όταν βλέπουμε ότι συστηματικά υπάρχει ανισότητα εις βάρος ε, κάποιων χωρών. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σε τρόπο. Και από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από, για το, από το 2004 ήταν μια αύξηση για τη χώρα μας 3%. Ας περάσουμε στο greening, το πρασίνισμα Κατανοούμε όλη την ανάγκη και τα προτερήματα να προχωρήσουμε προς αυτή την πορεία του πρασινίσματος. Είναι όμως αναγκαίο να είναι επαρκής στις ανάγκες των κρατών μελών αυτές οι προτάσεις και αυτά τα μέτρα και πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για το, ε, για το πρασίνισμα όπως η άρδευση και δεν βλέπουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ. Αντίθετα, είναι ε, μέτρα που εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τι χώρε του Βορρά, τι πιο πλούσιε χώρε και όχι τι χώρε του Νότου οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν συμπεριλαμβάνονται προτάσει για αυτό το πρασίνισμα για τι χώρε του Νότου. Εφισώ την προσοχή στι περιοχέ, στι χώρε του Νότου, ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση του προβλήματο τη απερίμωση που χρειαζόμαστε την άρδευση δεν είναι μόνο το, είναι πολλές φορές ε, η διάθεση νερού, ή ε, πολλές φορές ε, έχουμε και την προσαγωγή θρεπτικών ουσιών με αυτόν τον τρόπο στις καλλιέργειες οποροκυπευτικών και λαχανικών μέσω αυτής της άρδευσης. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις δυνατότητες. Και εδώ έχουμε και την κλιμακούμενη εφαρμογή. Τελικά πώς έχουμε μια πρόταση που επιτρέπει από το δεύτερο προς τον, πρώτο πυλώνα να σημειωθεί αύξηση, αλλά από τον πρώτο προς τον δεύτερο πυλώνα να έχουμε μόνο 10%. Αυτές είναι οι ασυμβατότητες ε, και που μας κάνουν να δυσπιστούμε για αυτή την πρόταση. Αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα. Ότι σε σχέση με ένα κράτος μέλος ε, ανακατανομή 40% των άμεσων επιδοτήσεων μέχρι το 2014 όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλέψει μέχρι, ε, σύγκληση μέχρι το 2029 η ε, ομοιομορφία των κριτηρίων και η δικαιοσύνη των κριτηρίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση. Αλλιώς θα έχουμε μεταρρύθμιση που θα είναι ψευδεπίγραφη, μόνο κατόνομα μεταρρύθμιση και σε σχέση με τον στόχο να είναι αυτάρκηση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα τρόφιμα και την, τον ανταγωνισμό της με, άλλα, με άλλες ε, υπήρους δεν θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση. Μάρτιν και μετά <clears throat> Είχα και εγώ κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να διατυπώσω. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να ξέρουμε πώς ε, αντλήθηκαν σημειώθηκε συνέχεια μιας ολόκληρης εξέλιξης και πήραν κάποιους συντελεστής εκ των έξω το θέμα των βιοκαυσίμων για παράδειγμα με την καλλιέργεια αραβοσίτου και αυτό είναι μια εξέλιξη που με άλλους τομείς ε, πολιτικών σημαντικά επηρεάζουμε και συνεπηρεάζονται. Δεν επιβάλλεται από κάποιους. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική αυτή που δίνει αυτά τα στοιχεία και πορεύεται με αυτόν τον τρόπο. Το άλλο θέμα είναι ότι μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη και μόνο μέσω της ε, ε, μεταρρύθμισης ε, στο σύστημα εκτατικής καλλιέργειας υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσο αφορά τα κράτη-μέλη. Σημαντικό θα ήταν να έχουμε και αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας τι γίνεται σε σχέση με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά, δεν αμβάνονται υπόψη με εξέπληξε ότι γίνεται λόγος και για αγρανάπαυση, για πάυση καλλιέργειας για κάποιες εκτάσεις. Έμαθα μέχρι σήμερα και το εκπροσωπούσα προς τα έξω ότι αυτές πρέπει να είναι οικολογικές ε, ε, κινήσεις. Πώς έχουμε τώρα πάλι την έννοια της αγρανάπαυσης που επανεισφραίει εδώ και σε σχέση με την Επιτροπή με μια άλλη αλληλουχία, μια άλλη σειρά ακολουθούνται τα πράγματα. Τώρα όμως αναφέρεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ανταγωνιστικότητα τι είναι, μια πολιτική που στοχεύει αποκλειστικά στις παγκόσμιες αγορές. Δεν μπορούμε άλλες πολιτικές και πολιτικούς στόχους να έχουμε μπροστά μας με τη μεταρρύθμιση που θα είναι πιο σημαντική για μας. Εσείς κλασικά πάλι θέτετε στο προσκήνιο ως στόχους αυτά που ουσιαστικά με την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν αλλά δεν μπορούν να είναι το κέριο κεντρικό σημείο της πολιτικής μας δράσης. Μεγκίνες. Καλώς. Μαγκίνες. Και μετά Μπρίτα Ρέμερ. Κύριε Μαγκίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λεπτομερή παρουσίαση. Διάβασα και εγώ το κείμενο που αφορούσε τις διάφορες παραγράφους και νομίζω ότι είναι μόνο το ανοιχτό τμήμα της συζήτησης. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειε και σαν οικονομολόγος υπεύθυνη γνώση των αγροτικών είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να δω όμως ποιος είναι ο αντίκτυπος σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Χαίρομαι για εξολόγηση αντικτύπου στο κείμενο αναφέρεται στη μείωση του περιθωρίου για τους ε, γεωργούς ε, και το κόστος ρόν αυξάνεται αλλά και οι τιμές των προϊόντων και προ, Προσπαθούμε να υπάρχει υποστήριξη εισοδήματο μέσω των άμεσων πληρωμών, ένα είδο υποστήριξη. Το παράρτημα 2 και εθνικέ οροφέ. Εκεί έχω ένα ερώτημα. Κάποιοι συνάδελφοι από την Πορτογαλία, τη Λετωνία και από αλλού το έθεσαν, και από τη Ρουμανία, ναι. Και ποιο ο ρόλο του Κοινοβουλίου, διότι θεωρώ ότι ε, σε κατεξιδότηση πράξη έχουν μείνει πολλέ λεπτομέρειε όσον αφορά τι άμεσε πληρωμέ και θέλω κάποιε διευκρινήσει. Δηλαδή, πώς έχει ειδικό ιδιαίτερο ρόλο το Κοινοβούλιο να παίξει, όχι μόνο όσον αφορά την αναδιανομή μεταξύ κρατών μελών, αλλά και εντός κρατών μελών. Ε, είναι σημαντική πτυχή αυτή. Από την εξολόγηση αντικτύπου φαίνεται ότι αν θέλαμε να είμαστε ειλικρινεί όσον αφορά το τομέα τη γεωργία, δεν θα θέλαμε να περιοριστούμε στον υφιστάμενο προπολογισμό, διότι προσπαθούμε να κάνουν πολλά περισσότερα οι γεωργοί όσον αφορά τα περιβαλλοντικά μέτρα παραδεχόμενοι όμως ότι η αγορά δεν τους πληρώνει και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ίδιους πόρους και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σω αυτό μπορεί να το σχολιάσει. Δηλαδή πόσο πραγματικό μπορεί να είναι αυτό, πόσο πραγματιστικό. Και να προσθέσω στι ανησυχίε που εξέφρασαν και άλλοι όσον αφορά τι λεπτομέρειε για το πρασίνισμα. Έκανα σχόλια προηγουμένω στη δική μου χώρα μέλο. Δεν θα είναι μεγάλο το ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εκεί που θα πρέπει να προσέξουμε κάτι είναι το εξή και ιδιαίτερα στην Επιτροπή μα οι έλεγχοι που αφορούν πολλές από αυτές τις προτάσεις. Συνάντησα κάποιες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Έχω τεράστιες ανησυχίες όσον αφορά τον ρόλο των ελεγκτικών φορέων, πώς κινούνται, πώς λειτουργούν και η μυστικότητα της διαδικασίας. Δεν την γνωρίζουμε μέχρι ότου περατωθεί και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουμε κάπως καλύτερα διότι υποθέτουμε ότι η έλεγχη είναι εκτός της εντολής μας σχεδόν μέχρι ότου έχουμε κάποιο συμπέρασμα, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα μας αφορούν ως ευρωβουλευτές. Δηλαδή θέλουμε πιο διαφανή διαδικασία, η οποία θα μας επέτρεπε να δούμε πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία κατά τη διάρκεια κάθε φάσεως, όχι μόνο όσον αφορά το τελικό πόρισμα, διότι ότι δρομολογηθεί ήδη ασκούμενες, ε, ασκούμενοι έλεγχοι αφορούν το 2006 κάποια κράτη-μέλη δεν έχουμε συντονιστεί ακόμα. Από αυτά που έχω ακούσει και βλέποντας το έγγραφο όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές βλέπω ότι θα αυξηθεί τελικά η γραφειοκρατία ε, και θα αυξηθεί και ο αριθμός των απαιτουμένων ελέγχων και θα αυξηθεί και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και είμαι κάθετα αντίθετη σε αυτό και θα έχω αντίρρηση, θα προβάλλω αντίρρηση σε κάθε στάδιο μέχρι ότου να το παραδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ένα πραγματικό και σοβαρό πρόβλημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες, Μπρίτα Ρέιμερς και μετά καλύνεται. Ευχαριστώ. Δύο μικρά σημεία θα ήθελα μόνο να αναφέρω και έχω ερωτήσεις για το πρασίνισμα, το greening. Όταν μελετήσατε τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, υπολογίσατε την άρνηση ε, των αγροτών, λίγοι ή πολλοί γεωργοί μπορούν να το αρνηθούν είτε γιατί δεν τους βοηθάει στην ανταγωνιστικότητα ή στη γραφειοκρατία. Και το δεύτερο, πώς υπολογίσατε το κόστος του πρασινίσματος και πώς ε, <clears throat> υπολογίζετε τις απώλειες εισοδήματος τι έχετε υπολογίσει. Γιατί οι αγρότε μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά από ό,τι εμεί στην πολιτική συζήτηση. Αυτά. Ευχαριστώ. Καλνιέται και Γιάρη είναι οι δύο επόμενοι θα πάρω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ όπως και οι προηγούμενοι να πω ότι βλέποντας την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Ιουνίου ε, εξεπλάγει. Διότι εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας εργαστήκαμε πολύ σκληρά για τις ε, πολιτικές κατευθυντικές γραμμές ε, και υιοθετήσαμε δύο ψηφίσματα. Μπορέσαμε να πετύχουμε κάποιο επίπεδο συμβιβασμών που ήταν κάτι αποδεκτό σαν αποτέλεσμα σχεδόν για όλα τα μέλη ε, της Επιτροπής. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου τι ήταν σημαντικό για τη χώρα μου και πιστεύω και για πολλές άλλες χώρες. Πρώτα απ' όλα, η αρχή της δικαιοσύνης όσον αφορά την διανομή, την κατανομή των άμεσων πληρωμών και άλλων οικονομικών πόρων για την γεωργία. Δεύτερον, συμφωνήθηκε ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εδράζεται επί αντικειμενικών κριτηρίων, όχι επί κάποιων συγκεκριμένων χρηματικών ποσών όπου προσαρμόζεται από αυτού του ποσού ένας τύπος για την κατανομή των πόρων, ε, καλύπτοντας διάφορες ανάγκες. Και τρίτον, υπήρξε συμφωνία επίσης ότι θα υπήρχε μια, ένα εύλογο μεταβατικό στάδιο, μεταβατικό διάστημα. Αυτή είναι μια διατύπωση που χρησιμοποιούμε για όλους. Γι' αυτό θα ήθελα να θέσω διάφορα ερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τις άμεσες ε, πληρωμές όταν τα νέα κράτη-μέλη προσχώρησαν στην Ένωση, όταν πραγματικά υποχρεωθήκαμε να αποδεχθούμε την πρόταση που έγινε βάσει της αρχής ότι ήταν η μοναδική επιλογή, λάβαμε τις άμεσες πληρωμές που σταδιακά α, έπρεπε να ενταχθούν μέχρι το 2013. Βασίστηκαν στην ιστορική αναφορά αυτές οι πληρωμές. Χρονολογεί το αυτή, αυτό το επίπεδο αναφορά στα μέσα τη δεκαετία του 90. Με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν η κατανομή των πόρων γίνεται βάση των ίδιων ιστορικών στοιχείων και προσαρμόζοντάς τα αυτά μόνο, αυτό για μένα είναι εντελώ απαράδεκτο, διότι τώρα, 20 χρόνια μετά και ίσως και 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχου του Βερολίνου, ακόμα χρησιμοποιούμε τι ίδιε αναφορέ για να προσαρμόσουμε τα, τις σύγχρονες ευρωπαϊκές γεωργικές πολιτικές. Λοιπόν, εξεπλάγει τα μάλλα όταν έμαθα ότι η χώρα μου, η Λετωνία, θα λάβει σε άμεσες πληρωμές το 2020 περίπου 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και δεν μπορώ να το εξηγήσω στον κόσμο στην Λετωνία. Κανείς δεν το δέχεται. Το ερώτημά μου είναι, γιατί μια άλλη αρχή που συμπεριλήφθη στο ψήφισμα που είχαμε υφετήσει στην Επιτροπή Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να υπάρχει οροφή και κατόφλιο για το μέσο όρο για οποιονδήποτε γεωργό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η εξολόγηση αντικτύπου για αυτό το περιθώριο από 120% με 80% ανακτάριο. Στην περίπτωση της Λετωνίας υπολογίσαμε ότι αυτά αφορά 7 χρόνια περίπου, για 7 χρόνια περίπου 700 εκατομμύρια. Λίγα χρήματα που χρειάζονται για να υπάρξει δικαιοσύνη και ισοτιμία όσον αφορά την αγροτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση η οποία ήδη τη στιγμή που ανακοινώθηκε, τη στιγμή θα ανακοινωθεί, θα δημιουργήσει ένα νέο κύμα διαπραγματεύσεων για την επόμενη μεταρρύθμιση. Θα πρέπει αυτή τη φορά να κάνουμε μια καλή μεταρρύθμιση που θα είναι αποδεκτή για τους γεωργούς μας, αλλά αποδεκτή και για το ευρύτερο κοινό, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Γεωργία να γίνει ισχυρή, ανταγωνιστική το παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κανιέτε. Γιάρ και Κώστιγκερ είναι οι επόμενοι δύο μιλητέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις έχω εγώ στην τοποθέτηση του κυρίου Χανιώτη. Πρώτον, για τον προπολογισμό. Γιατί στο μεταξύ η ερώτηση είναι πόσα λεφτά έχουμε και στο μεταξύ κυκλοφορούν τρία διαφορετικά ποσά. Το ένα είναι από τα κράτη-μέλη, το άλλο από την Επιτροπή Γεωργίας και το ε, επόμενο από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Από ποιον προϋπολογισμό λοιπόν ε, ε, ξεκινάτε για τους προϋπολογισμούς σας. Για τις άμεσες πληρωμές τώρα. Πόρτα η προσαρμογή ή ε, η συμπλησίαση. Πώς να το πω, αυτό τυχαία το υπολογίζεται. Υπάρχει καμιά συγκεκριμένη αρχή, καμιά μαθηματική αρχή, ένας μαθηματικός τύπος, για να υπάρχει και μία περατότητα. Δηλαδή ας πούμε ότι έχει ένα χ κόστος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενιαίο παντού το ίδιο ή συγκρίσιμο, ε, ο τελικός στόχος ποιος θα είναι για να καταλάβουν και τα κράτη που είναι κάτω του μέσου όρου στις άμεσες πληρωμές. Ε, θα επιθυμούσα να έχω έτσι μια ε, πιο επιστημονική βάση για να στηρίξω τις αποφάσεις μου. Τρίτη ερώτηση, το πρασίνισμα και το κόστος. Σε μία παρενθετική πρόταση είπατε ότι για τις ε, εκμεταλλεύσεις που ήδη πληρούν κάποιες προϋποθέσεις πρασινίσματος ισχύουν τα εξή. Αυτό τι σημαίνει. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν ήδη κάποιες εκμεταλλεύσεις ε, που πληρούν τα κριτήρια. Γι' αυτό έρχομαι στην τέταρτη ερώτηση. Τότε γιατί τους επιβαρύνουμε με έξτρα γραφειοκρατία. Δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα δεν θα μπορέσουν να αποδεσμευτούν από ε, το ζήτημα αυτό της υποχρέωσης του ε, πρασινίσματος. Και τελευταία ερώτηση για το Small Business Act. Μας δώσατε πολλά παραδείγματα και υπάρχουν και αντίστοιχα και για τη Γερμανία. Εγώ θεωρούσα ότι αυτή η πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις είναι ένα θέμα εθελοντικό. Δηλαδή, ε, μπορεί κάποια κράτη να μην ποντάρουν σε αυτό το χαρτί να μην το παίξουν αυτό το χαρτί. Λάθος το κατάλαβα, δεν είναι εθελοντικό, είναι υποχρεωτικό αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κέστιγκερ. Και μετά ο Αντιπρόεδρος Βατσιόσκι. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Στην αρχή αναφερθήκατε ε, στην παραγωγή ζαχάρεως και τονίσατε ότι έχετε υπολογίσει ότι και στο μέλλον στη Βραζιλία θα είναι αυξημένη η παραγωγή βιοεθανόλης. Τώρα έχουμε την πρόταση που λέει ότι το 2015 θα καταργηθεί η ποτόστοση αυτή ένα χρόνο νωρίτερα. Ε, σήμερα στην Ευρώπη όμως μπορούμε να εξασφαλίσουμε μόνο το 85% των αναγκών μας. Έχουν ε, κάνει υπολογισμούς οι υπηρεσίες σας ε, σε περίπτωση που πέσουν οι παγκόσμιες τιμέ, τι θα γίνει, ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσει αυτά τα φαινόμενα και ποιε απαντήσεις δίνουμε στους παραγωγούς για την ασφάλεια τροφίμων. Γιατί και η Ευρώπη είναι ένας τόπος παραγωγής ε, εγγυημένη και οι ποσοστώσεις ε, μου φαίνεται καλό μέσο παραγωγής γιατί είναι και ένα στοιχείο που μπορούν να κανονίσουν την πορεία τους οι παραγωγοί. Και οι γεωργοί δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν ε, προϊόν, καλλιέργεια. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ελάχιστη ασφάλεια προγραμματισμού. Μια άλλη ερώτηση αφορά το πρασίνισμα. Εκεί έχετε στοιχεία αριθμητικά για τον πρώτο πυλώνα. Τι θα σημαίνει για τα κρατη Στο δεύτερο πυλώνα ε, γίνονται ήδη πολλά στα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για το περιβάλλον. Έχετε κάνει υπολογισμούς όλα αυτά τα κράτη πώς θα τα μεταφράσουν στον πρώτο πυλώνα, γιατί όλα αυτά τα υποχρεωτικά νέα μέτρα, τα τρία που προτείνετε, μπορεί να είναι κάτι που θα φέρει σε μειονεκτική θέση ορισμένες εκμεταλλεύσεις. Έχετε υπολογίσει εκεί, έχετε αριθμητικά στοιχεία και σε σχέση με τόσα είπε η κυρία Μαγκίνες, πραγματικά εμείς υπολογίζουμε το διοικητικό κόστος και το κόστος του ελέγχου να αυξηθεί και με αυτά τα μέτρα για το πρασίνισμα. Αυτά τα έχετε εκτιμήσει, έχετε δει τι σημαίνει αυτό ως διοικητικός φόρτος και γραφειοκρατικό κόστος για το έλεγχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κόσιγκερ. Αντιπρόεδρος Βασεκόφσκι και μετά ο Τζόρτζ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω ότι συμφωνώ πλήρως και απόλυτα με αυτά τα οποία ο κύριος ε, Νικουλέσκου από πλευρά κυρία Κονιέτα και για, από άλλους για την αδικία του καθεστώτος των άμεσων πληρωμών. Έχω κάνει λόγο επανειλημμένα και πολλές φορές στα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής για αυτό το θέμα και έτσι δεν θα επαναλάβω τις θέσεις μου. Θα θέλω όμως να τονίσω από την άλλη πλευρά ότι είναι απαράδεκτο για μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε εμείς οι ευρωβουλευτές από χώρες που βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση και είναι σαφές αυτό, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες προτάσεις. Πώς θα μπορούσαμε ως αιρετοί εκπρόσωποι των κοινωνιών μας να έχουμε καθαρό το μέτωπο αν συμφωνήσουμε με τέτοιες προτάσεις. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την ανατροπή της ΚΑΠ και έναντι των αρχών που, ε, επί των οποίων βασίζεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την ε, ψευδεπίγραφη κατάσταση όπου δεν υπάρχει δικαιοσύνη και επικρατεί αδικία, όπου χώρες όπου έχουν πιο μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, εκεί παίρνουν μεγαλύτερη υποστήριξη οι γεωργοί από ό,τι σε χώρες που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη και δυσμενέστερη θέση. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με μια τέτοια φιλοσοφική προσέγγιση. Εκείνοι που είχαν πολλά στο παρελθόν να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα, εκείνοι που είχαν λίγα να γίνουν ακόμα φτωχότεροι και να μην έχουν τίποτα. Αυτό θα σήμαινε να προσυπογράψουμε την αρχή της αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει αυτές τις διαφορές και τις ανισότητες, να μην υπάρχουν χασμα, ε, κενά και διαφορές ε, μεταξύ των ε, χωρών να λάβετε υπόψη ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τα νέα κράτη-μέλη και δεν έχει γίνει για παράδειγμα λόγος για αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν χώρες όπου η, η γεωργία πραγματικά χάνει τον ρυθμό της και φθήνει και χάνει την ζωτικότητά της ενώ χρειάζεται μια ισχυρή γεωργία η Ευρώπη πανευρωπαϊκά, πανενωσιακά. Αυτή η πρόταση του 1 τρίτου μέχρι 90% του μέσου όρου πώς να το πω, και αυτό είναι πάλι μια αρνητική διακριτική μεταχείριση. Δεν είναι ότι θα φτάσουμε μέχρι το μέσο όρο. Τώρα ακούμε μέχρι 90% λέει ε, θα μπορούμε να φτάσουμε και ένα τρίτο θα είναι το αντίστοιχο που θα παίρνουμε. Και αυτό δεν έχει καμιά λογική και είμαστε οι υπεύθυνοι αιρετοί εκπρόσωποι των ψηφοφόρων, των πολιτών μας. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες προτάσεις. Προσδοκούμε και προσβλέπουμε σε μια δίκαια πρόταση, ισοδίκαια, που θα βασίζεται σε αντικειμενικά αμερόληπτα κριτήρια. Πρέπει όλες αυτές οι προτάσεις, αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Ευχαριστώ Τζος Λάιν και μετά Τζιμ Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Τάσο Χανιώτη για την παρουσίασή του. Έχω τέσσερα σημεία τα οποία θέλω να θίξω. Τώρα όσον αφορά την, ε, το μοντέλο κατανομής ε, που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να εξηγήσετε γιατί χρησιμοποίησατε το μοντέλο που κάνει τη μικρότερη αναδιανομή, ανακατανομή. Γιατί διαλέξατε το μοντέλο που λέτε ότι κλείνεται μόνο των τρίτων του, της διαφοράς, γιατί όχι 50%. Γιατί όχι τουλάχιστον ε, μια ελάχιστη πληρωμή ανακτάριο που ισοδυναμεί με 75% διότι αυτό συζητήθηκε. Όταν κάνετε εξολόγηση αντικτύπου να εξηγήσετε γιατί διαλέξατε την ελάχιστη ε, ανακατανομή που ήταν εφικτή βλέποντας τις προτάσεις που κάνατε. Δεύτερον, όσον αφορά τα μέτρα για το πρασίνισμα, αναφερθήκατε στην πράσινη κάλυψη. Βλέποντας λοιπόν τις προτάσεις σχετικές, ε, καλύπτει πάρα πολλά τετραγωνίδια όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Ε, τι πρόβλημα ελέγχου δημιουργείται. Τι σας υποχρέωσε ή σας έκανε να μην επιλέξετε αυτή τη δυνατότητα όσον αφορά την πρόταση για το πρασίνισμα. Μετά, που έγκυται, εδώ μάλλον που μας ανησυχεί, όπου εμφανίζεται η πραγματική γραφειοκρατία. Μιλώντας σε κάποιες αρμόδιες αρχές και σε άλλους, εξέφρασαν ανησυχίες. Δηλαδή τις προτάσεις ε, για, που δίνονται για τον πραγματικό Γεωργό. Και συμπλήρωση εισοδήματο. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα με την γραφειοκρατία για την εφαρμογή. Για τον ενεργό αγρότη. Όταν απαιτείται τζίρος τουλάχιστον 5% από τη γεωργία. Γεωργικός τζίρος πώς καθορίζεται. Πώς εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν, που έχουν χωριστεί στα δύο για να γίνουν επιλέξιμες. Πώς μπορείτε να επιλέξετε την, το γνήσιο διαχωρισμό και το διαχωρισμό που γίνεται για να ξεγελαστεί η νομοθεσία. Μπορείτε να εξηγήσετε πώς οι αρμόδιες αρχές τα, τα κρίνουν όλα αυτά. Τι πληροφορίες θα απαιτηθούν Μετά, δεύτερον, η προτάσή σας για, για το συμπλήρωμα εισοδήματος. Βλέπω τη συγχρολόγηση που κάνατε. Και η πρόταση λοιπόν αυτή για τη συμπλήρωση του δήματος είναι πάρα πολύ μικρή χαμηλή όσον αφορά τα χρήματα που παράγει τελικά. Άρα ερώτημα, πώς το καλό αυτή η πρόταση θα λειτουργήσει, λαμβάνοντας υπόψη θα χρησιμοποιήσετε ε, κάποιες μονάδες εργασίας για να δείτε κατά πόσο έχουν ξεπεράσει τα νότατα όρια οι γεωργοί. Πώς θα κρίνετε ποιος είναι ο καλή τυπίστη πραγματικός Γιωργός ε, ή κάποιος που εφευρίσκει τη θέση. Ε, οι συγγενείς που εργάζονται είναι πραγματικά εργαζόμενοι, αποτελούν μέλος επιχείρησης, άρα δεν είναι απασχολούμενοι από την επιχείρηση πραγματικά. Υπάλληλοι αν θέλετε. Και ποιο είναι το χρηματικό όριο, διότι έχουμε 27 διαφορετικές χώρες με διαφορετικά επίπεδα αμοιβών για τους εργαζομένους. Πώς αποφασίσετε πιο δεδειγμένο επίπεδο ε, αμοιβή. Θα καθοριστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματο, θα υπάρχουν 27 διαφορετικά επίπεδα εισοδημάτων ανάλογα με τι διάφορε χώρε. Εδώ έγκυται η πραγματική γραφειοκρατία και θα ήθελα κάποιε εξηγήσει όσον αφορά τη σκέψη που ε, κρύβεται πίσω από το πώ θα εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχέ κάποιε από τι προτάσει και κυρίω αυτό το συμπλήρωμα του εισοδήματος που παράγει ε, σχεδόν ελάχιστα μηδενικά ποσά για να μεταφερθούν στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ, George. Τζίμι Νίκολσον και μετά ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ο Τζίμι είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χανιώτη για την εξαιρετική παρουσίαση. Έχω την αίσθηση ότι ε, ίσως μας λένε ε, αυτά που θέλουμε να ακούσουμε ε, ε, και όχι να δούμε την πραγματικότητα όπως έχει. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε εδώ, ζούμε σε ένα κόσμο πάρα πολύ ασταθή και αγορές πάρα πολύ ασταθείς. Σε έξι μήνες μπορεί να έχει αλλάξει ριζικά η κατάσταση και τότε τι θα γίνει. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα πρέπει τακτικά να προσπαθούμε και να προσαρμοζόμαστε. Έχω πολλές ανησυχίες εγώ για όλη αυτή την κατάσταση και πολλές επίσης σε σχέση με αυτά που είπαν και ο Τζόρτζ και η του Μαγκίνες. Πολλά από αυτά τα θέματα στη Γεωργία όπως και αλλού στην Ευρώπη, ε, στις οδηγίες, αλλά είναι πώς εφαρμόζεται η οδηγία σε επίπεδο κράτους μέλους και τι ερμηνεία δίδεται, όχι η ίδια η οδηγία, αλλά πώς τα ερμηνεύουν αυτά τα κράτη. Γι' αυτό έχουμε τόσες διαφορές ενδεχομένως για μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Πόσο περισσότερη γραφειοκρατία και χαρτομάνη θα ε, προσθέσει αυτό το πρασίνισμα. Πόσες περισσότερες επιθεωρήσεις θα γίνονται στις εκμεταλλεύσεις ε, και τι θα δουν οι γεωργοί να τους επιβαρύνει. Γνωρίζουμε όλη την πολλαπλή συμμόρφωση, το cross compliance. Αυτό ε, πόσα περισσότερα χρήματα θα σημάνει. Όταν αρχίζουν οι ελεγκτές και οι λογιστές να ελέγχουν το μέλλον της γεωργίας, θα πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε γιατί στη μικρή μου χώρα που ονομάζεται Βόρεια Ιρλανδία, έχουμε περίπου 100 εκατομμύρια σε ε, στα χαρτιά, αλλά το θέμα είναι πώς τα ερμηνεύουν οι λογιστές, οι ελεγκτές και πού είναι αυτά τα 100 εκατομμύρια. Και δεν μπορούμε να τα επομιστούμε. Αυτά όλα τα βρίσκω απαράδεκτα. Τι κάνουμε λοιπόν για το πρασίνισμα. Θέλω να ξέρω τι σημαίνει αυτό για τους γεωργούς, πόσο θα τους επιβαρύνει. Και έχουμε την ευκαιρία τώρα ε, να δούμε το μεγαλύτερο γραφειοκρατικό εφιάλτη που έχει δει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα αυξήσει και το κόστος ε, και της γραφειοκρατίας και της διοικητική δουλειά και του χαρτοβασιλείου και ε, δεν θα κάνουν άλλη δουλειά από το να συμπληρώνουν έγγραφα οι γεωργοί αντί να καλλιεργούν και να παράγουν τρόφιμα. Τελικά εκεί θα καταντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα κάνω μια πολιτική αξιολόγηση της τεχνικής δουλειάς που παρουσιάστηκε, διότι η πολιτική μας εταίρη δεν είναι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είναι η ίδια Επιτροπή και ο Επίτροπος. Εν πάση περιπτώσει, χαιρετίζω και ευχαριστώ για το έργο, την εργασία που παρουσιάστηκε και σε σχέση με, τις, ε, με την πρόταση που ε, έγιναν δείχνουν ποιε είναι οι κατευθύνσει και οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν είναι οι δικέ μα και πρέπει να βελτιώσουμε αυτέ τι προτάσει ώστε να υπάρξει πλειοψηφία και να μπορέσουμε να πορευτούμε προ τη σωστή κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αν θα θυμόσαστε η έκθεση DES ήταν εκείνη στην οποία προτείναμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ελάχιστο ε, κατόφλι στο οποίο θα έπρεπε να τίνουν τα κράτη-μέλη. Αλλά εγκρίναμε επίσης ότι θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ανώτατο ανόφλι, ανώτατο ανόφλι, ώστε να βρισκόμαστε μέσα στο κεκτημένο, στη σωστή πορεία. Και βλέπουμε από το γράφημα σε σχέση με τη μελέτη των επιπτώσεων που ε, έχουμε ως προοπτική, οι τεχνικοί είχαν την προσοχή να θέσουν το 90% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξέρω, μια και υπάρχει απουσία κάποιας γραμμής πάνω από το 100% μέχρι το 100% αυτό είναι, α, ας το πω έτσι, παράληψη ή ήταν ε, εσκεμμένο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα όσα είχε προτείνει στην έκθεση ΝΤΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε με τη σειρά μου. Όπως και οι συνάδελφοι θέλω να πω ότι συμφωνώ ότι είναι μια καλή αυτή η παρουσίαση που έγινε αλλά δοθέντων των όσων είπαν οι συνάδελφοί μου, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονται καθόλου στις προσδοκίε μα, στι προσδοκίε των κρατών μελών. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία. Πιστεύω ότι η κατανομή του 1 τρίτου τη διαφορά του 90% του μέσου όρου του ευρωπαϊκού των αμέσων πληρωμών από την αρχή θέτει το επίπεδο των πληρωμών κάτω από το μέσο όρο και νομίζω ότι αυτό είναι ανεπαρκέστατο. Πιστεύω ότι κάποιες χώρες, όπως είναι η χώρα μου, η Ρουμανία, θα φτάσουν στο 100% των πληρωμών το 2016. Είναι σαν να ξεκινήσουμε για κάποιο ταξίδι υπό τους ίδιους όρους, αλλά κάπου στο δρόμο αλλάζουν οι όροι. Και είναι προφανές ότι λείπει κάποια ισοτιμία όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρομοίως, θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο η πράσινη διάσταση θα εφαρμοστεί, το πρασίνισμα, στη Γεωργία. Διότι σε αυτές τις συνθήκες κινδυνεύουμε να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Δοθέτω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μόνο 6% των γεωργών είναι νέοι και 2 τρίτα ανήκουν στη γενιά που είναι πάνω από 55 ετών, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας φαίνεται δίκιο να έχουμε μόνο 2% των πόρων που διατίθεται για κάθε κράτος μέλος ώστε να υποστηρίξουν τους νέους ε, γεωργούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλμπερντές και μετά κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή για την εισήγηση, την παρουσίασή του στην Γερμανία. Έχουμε μια παροιμία που λέει Εβεί έτεινα και πρέπει με πίστη να ακούσω και να υλοποιήσω. Εδώ άκουσα όμως τα όσα είπατε, τα λόγια, αλλά τη λογική δεν μπορώ να κατανοήσω απόλυτα. Και παρότι προέρχομαι από την Γερμανία, υποστηρίζω την Σάντρα Κανιέτε και άλλους συναδέλφους και ε, ευρωβουλευτίνες και ευρωβουλευτές που άσκησαν επικρίσεις ε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν λαμβάνει υπόψη την ισόνομη και ισοδίκαιη κατανομή των κονδυλίων για την υποστήριξη στην Ευρώπη. Εδώ πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αν δω τους αριθμούς, για την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία, αν προσθέσουμε πρώτο και δεύτερο πυλώνα, 332 ε, ευρώ βρίσκεται σε σχέση με τον ε, μέσο όρο. Όμως, ε, όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, βρίσκεται πολύ πίσω η Πορτογαλία. Θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόταση της Επιτροπής, ώστε τα κράτη-μέλη που βρίσκονται πολύ κάτω από το μέσο όρο να παίρνουν περισσότερα χρήματα από το δεύτερο πυλώνα που θα μεταθέτουν, μετατίθενται στον πρώτο πυλώνα, ώστε να μπορέσουν αυτές οι αδικίες να αμβληθούν και να εξισορροπηθούν και συγχρηματοδότηση που πρέπει να υπάρχει από το δεύτερο για το δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Εδώ πρέπει να κάνει τη δουλειά της σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί διαφορετικά σύμφωνα με συνθήκες Λισαβόνας εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο θα υποβάλουμε προτάσεις προς βελτίωση, τροποποίηση αυτών των προτάσεων με βάση τη συνθήκη τη Σαββόνα. Εκείνο το οποίο με εξόριξε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν έχω υπόψη τον Επίτροπο για τη Γεωργία αλλά άλλου επιτρόπου επίση ότι κάποιες σαφέστατες ενδείξεις ε, της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της έκθεσης ΔΕΣ δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη. Η παράταση της ε, ε, κοινή οργάνωσης αγοράς για τη ζάχαρη μέχρι το 2020 θεωρούμε ότι αυτό δεν ήταν σωστό από πλευράς της Επιτροπής να μην ληφθεί αυτό υπόψη. Και όσον αφορά και τον Ίνο και πάλι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άκουσε, δεν έτεινε βίκο νου στι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω τι γίνεται εδώ. Διότι βλέπουμε ότι παρακάμπτει πλήρω ε, τι προτάσει του Ευρωκοινοβουλίου η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που εμένα και του γεωργού που εκπροσωπώ και πολλού συναδέλφου εδώ μα ανησυχεί όλου είναι το γεγονό ότι αυτέ οι προτάσει ιδιαίτερα αναπόφευκτα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρηση. Θα ήθελα να μου πείτε, να ξέρω αληθεύει, ακούμε φήμε ότι ακόμα λέει και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκινείται από κάποιες υποθέσεις ότι τουλάχιστον 5% μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρηση θα προσκληθεί. Αν εν τη συνέση και σοφία της ε, επιφυλακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα υπάρξει 5% μεγαλύτερη επιβάρηση, τότε θα είναι 20% σίγουρα η ε, γραφειοκρατική επιβάρηση. Μετά το κόστος του πρασινίσματος, του greening. Αν δει κανείς ένα χίποσο ποσό, για παράδειγμα, για το πρασίνισμα, παράδειγμα, 40 50 ευρώ, ευρώ έστω. Ε, τότε θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και έντιμοι και να πούμε στους γεωργούς εκεί έξω ότι ακούστε οι αντισταθμιστικές πληρωμές θα μειωθούν κατά αυτό το ποσό χ ψ διότι όταν υπάρχουν δαπάνες ε, τότε αυτό τι θα σημαίνει μείωση λοιπόν των ποσών που θα παίρνουν οι γεωργοί. Πρέπει να το πούμε αυτό στους γεωργούς και προς το κοινό, προς τους πολίτες. Και εδώ κάτι άλλο που ε, θα ήθελα να προσθέσω σε επιπλέον παρατήρηση, αυτό το 5% συμμετοχή στο εισόδημα μπορεί ίσως να είναι μια καλή πρόθεση σε κάποιους μεγάλους εισοδηματίες ε, να τους αποκλείσουμε κάποιος που κερδίζει ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο για παράδειγμα. Αυτός δεν θα εξαρτάται από αντισταθμιστικές πληρωμές όμως, όμως με αυτό το γραφειοκρατικό 5% ως επιβάρηση ο στόχος της ισοδίκαιας ε, μεταχείρισης όσον αφορά τα υποφορβία και την κτηνοτροφία μικρών ε, εκμεταλλεύσεων και μονάδων που έχουν άλογα και εκτρέφουν άλογα δεν μπορεί να ε, δικαιώσει καθόλου αυτούς τους ανθρώπους. Οδηγεί σε μαζική γραφειοκρατική επιβάρηση για πάρα πολλούς γεωργούς και στο τέλος ε, θα πρέπει να υποβάλλονται πόσα στοιχεία για να αποδειχθεί ότι αυτό δεν ισχύει για αυτούς. Βλέπω λοιπόν ότι δεν θα είναι λειτουργικά όλα αυτά και θα έχει πολλή δουλειά το Κοινοβούλιο να τα βελτιώσει τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ αγαπητέ Άλμπερτ. Συγκεριέσκει και κλείνει, κλείνει γύρω παρεμβάσεων. Ευχαριστώ. Ε, αυτή είναι το πρώτο ερώτημα που έχω. Οι προτάσεις για τις μικρές εκμεταλλεύσεις πώς θα επηρεάσουν δομικές αλλαγές που θα χρειαστούν αυτές οι εκμεταλλεύσεις στα διάφορα κράτη-μέλη, μακροπρόθεσμα. Χτες, εννέα περιφέρειες από Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία υπέγραψαν μια κοινή θέση όσον αφορά την γεωργική πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου για τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Στις περιφέρειες λοιπόν αυτές, όπου οι δομές των εκμεταλλεύσεων είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένοι. Μόνο κριτήριο θα είναι η έκταση ή και ο αριθμός των εργαζομένων στις εκμεταλλεύσεις αυτές. Το ίδιο ισχύει και για εκμεταλλεύσεις σε ορεινέ περιοχές. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μεταφορές μεταξύ πυλώνων. Ποιε είναι οι συνέπειες των αλλαγών αυτών τη μετακινήσεω των πόρων. Δεν βλέπω σχετική ανάλυση στην παρουσίαση. Τρίτον, διατείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αντικειμενικά κριτήρια ανακατανομής θα εφαρμοστούν στο δεύτερο πυλώνα. Ερώτημά μου, αυτό γιατί δεν ισχύει για τον πρώτο πυλώνα. Και άλλο ένα ερώτημα. Στα πλαίσια του άρθρου 38, στήριξη με βάση την παραγωγή. Αυτό που λείπει είναι ο καπνός, ο τομέας του καπνού. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι ο καπνός καλλιεργείται από μικρές εκμεταλλεύσεις, είναι ένας τρόπος εξάλληψης της ανεργίας, μείωσης ανεργίας και η παραγωγή του καπνού δεν σχετίζεται καθόλου με την χρήση ε, των τσιγάρων από τους ε, πληθυσμούς των χωρών. Όσον αφορά το μέα της ζάχαρης, η αξιολόγηση συνεπειών αντικτύπου υποθέτει ότι το σενάριο χωρίς ποσοστώσεις, δηλαδή οι, οι εκτάσεις καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων, με καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων θα αυξηθεί. Πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα, σε αυτό το αποτέλεσμα. Παρόλο που θα μειωθούν οι τιμές δηλαδή, η έκταση όμως που, στις οποίες, ε, οι εκτάσεις στις οποίες θα καλλιεργείται το ζαχαρότευτο θα αυξηθούν. Και άλλο ερώτημα που αναφέρεται στη θέση που έχουν στην πολιτική συνοχή οι περιοχέ υπαίθρου, γιατί φαίνεται να το λησμονούμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Κύριε Σεγκερέσκη, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, και εγώ θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις πριν δώσω το λόγο εκ νέου στον Τάσο Χανιώτη και στους άλλους συναδέλφους της Γενικής Δευθύνσεως Γεωργίας. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια θέματα μεταξύ μας. Είναι σαφές, σαφής οι επικρίσεις. Υπάρχει και αρκετή ε, ε, ε, ταύτιση απόψεων σε αυτά που άκουσα. Λοιπόν, θα πρέπει να περάσουμε σε προτάσεις λόγω της συναπόφασης. Οπότε θα ήθελα να υπογραμμίσω στου εισηγητέ και στου σκιώδη εισηγητέ ότι φτάνει η στιγμή που θα πρέπει να κάνουμε κάποια συνθετική δουλειά μεταξύ μα, να αρχίσουμε να οικοδομούμε, να κατασκευάζουμε κάποια υπόθεση, κάποια σενάρια για να τα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήθελα όλοι να συνεχίσουμε αυτό το εγχείρημα κριτικής χωρίς να περάσουμε ταχύτερο δυνατόν σε μια ε, φάση που θα κάνουμε προτάσεις. Και μετά θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στον Τάσο είναι απαραίτητο το ταχύτερο δυνατό να έχουμε και το ε, κριτήριο κατανομής για το δεύτερο πυλώνα. Γιατί αφασβήτητα αν δεν έχουμε τα στοιχεία, αν δεν έχουμε τα ακριβή νούμερα, εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια απόσταση όλο και μεγαλύτερη μεταξύ των 12 νέων κρατών μελών που θα θέλουν, όπως επανειλημμένα υπογραμμίστηκε, να προχωρήσουν πιο γρήγορα και απ' την άλλη θα έχουμε την έλλειψη των και η έλλειψη πόρων δεν μα επιτρέπει να κινηθούμε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Άρα χρειάζεται να έχουμε ένα πλήρε πλαίσιο όσον αφορά την κατανομή μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα σε όλε τι χώρε. Πότε θα έχουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Πότε θα έχουμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ όλου. Λοιπόν, ο τάσο Χανιώτης έχει το λόγο. Δεν ξέρω ποιο θα πάρει το λόγο. Κανεί το Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τα σχόλια όχι μόνο είναι επικοδομητικά και χρήσιμα, αλλά είναι σχόλια που πρέπει πολύ σοβαρά να λάβουμε υπόψη σε σχέση με την προπαρασκευή αυτής της πρότασης. Να κάνω μια διαφοροποίηση και ο κύριος Καπόλα Σάντος ε, συνέφερε, συνεισέφερε σε αυτό. Είμαι εδώ παρόν για να παρουσιάσω το αναλυτικό πλαίσιο το, του πώς καταλήξαμε σε αυτές τις προτάσεις. Όπως ε, προανέφερα υπάρχουν αποφάσεις ε, που λαμβάνονται που βρίσκονται σε πολιτικό επίπεδο και είμαι βέβαιος ότι θα δοθούν αποσαφηνήσεις στο δεδομένο πολιτικό επίπεδο σε εσά. Ιστερότερα. Επειδή όμως πολλές ερωτήσεις ε, επικεντρώνονται στη δικαιοσύνη και στην κατανομή στον επιμερισμό της ε, δικαιοσύνης. Είναι σημαντικό να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Θα δείτε στη μελέτη επιπτώσεων και θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω για αυτό. Έχουμε διάφορα σενάρια, ιδιαίτερα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν για το flat rate, το 80%, το 100% και 120% και όλα αυτά τα ενδεχόμενα σενάρια. Αυτά είναι όλα διαθέσιμα και έχουν δημοσιευθεί. Όταν φτάνουμε όμως στο, στο, στο σημείο της κατανομής αυτής της βοήθειας. Ξεκινώντας με το θέμα της δικαιοσύνης, πρέπει ένα θεμελιώδες ερώτημα θεθεί. Δικαιοσύνη έναντι τίνος. Και για μας το πιο σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της πρότασής μας ήταν σε σχέση με τους στόχους που εμείς είχαμε θέσει και που θα έπρεπε να επιτευχθούν με τις άμεσες πληρωμές. Στο παρελθόν οι άμεσες πληρωμές καθοριζόντουσαν από την αρχή της υποστήριξης του εισοδήματος των γεωργών. Σήμερα καθορίζονται όλο και περισσότερο από την ανάγκη του να υπάρχει η κοινή προσπάθεια που πρέπει να υποστηριχθεί και οικονομικά και περιβαλλοντικά η προσπάθεια των γεωργών. Γι' αυτό έχουμε συνδυασμούς δύο ευραίων ομάδων κριτηρίων, οικονομικών κριτηρίων και περιβαλλοντικών κριτηρίων. Τούτων λεχθέντων το πρώτο θέμα το οποίο συνδέεται με τα οικονομικά κριτήρια είναι φυσικά το εισόδημα. Και είμαι σχεδόν βέβαιος πρέπει να πω ότι το επιχείρημα της δικαιοσύνης σε σχέση με τα κράτη-μέλη διαφορετικά αντιμετωπίζεται όταν έχουμε τη σύγκριση μισθών σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πράγμα το οποίο δεν θεωρούμε ότι πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στο ίδιο επίπεδο, εκτός αν υπάρχει μια συνολική πολιτική σύγκληση. Αυτά είναι τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Λαμβάνοντας αυτά τα κριτήρια, σε ένα ιδανικό κόσμο, οι τιμές θα έπρεπε να αντανακλούν την παραγωγικότητα και θα έπρεπε να μας δίνουν την καλύτερη, θα έλεγα, τον καλύτερο προσανατολισμό πώς θα έπρεπε να διαμορφώνεται η υποστήριξη. Όπως όμως είδαμε με μια ευρεία μελέτη, η κατάσταση όσον αφορά τις αγορές δεν είναι ούτε ιδανική ούτε τέλεια. Και τι κάναμε. Και θα ήθελα να το δούμε στην οθόνη, στη σειρά αυτή των γραφημάτων, των στοιχείων, των διαφορετικών κριτηρίων που χρησιμοποίησαμε. Λοιπόν, αυτό που θα δείτε στον πίνακα που θα προβληθεί ως γράφημα, τώρα στην οθόνη σε λίγο, μάλιστα, ειδού, ο πίνακας εμφανίζεται τώρα. Αυτό που έχουμε στην κάθετη, στον κάθετο άξονα και με πολύ μικρά γράμματα είναι τα διαφορετικά κράτη-μέλη και στο οριζόντιο επίπεδο τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε. Οικονομικά, αγοραστική δύναμη, ΑΕΠ, ανακεφαλή, ε, όσον αφορά τις, ε, την παραγωγικότητα ανά και την αντανάκλαση αυτών των στοιχείων. Και έχουμε και το ε, την έκταση που χρησιμοποιείται ως ποσοστό του συνολικού, της συνολικής επικράτειας, νατούρα ως έκταση σε εμβαδών, εκτάσεων και αυτό που θα ήθελα να κάνουμε είναι να ταυτοποιήσουμε για παράδειγμα ένα κράτος στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε και εδώ με δύο σταυρούς έχουμε τα πιο θετικά κριτήρια που μπορεί κανείς να δει που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος. Με ένα σταυρό Έχουμε κριτήρια θετικά, αλλά χαμηλότερης ε, ε, ε, εμβέλειας. Έχουμε αρνητικά με ένα πλήν, αρνητικά στοιχεία, με δύο πλήν, πολύ αρνητικά στοιχεία. Α, ταυτοποίηση λοιπόν αντικειμενικών κριτηρίων για τον επιμερισμό. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία άμεσα μπορεί να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα ότι εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί να ισχύει μια, ο κανόνας της δικαιοσύνη, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Θα δείτε την πραγματιστική προσέγγιση, ρεαλιστική προσέγγιση που προτείνουμε εμείς με αυτούς τους πίνακες που αντανακλά και την πραγματικότητα. Μετακινούμενοι δηλαδή προς ένα μεγαλύτερο βαθμό εναρμονισμού μεταξύ των κρατών μελών, όχι μόνο θα περιορίζεται η προσπάθεια από τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ε, ε, ε, κατανομή αλλά και από μεγαλύτερης εμβέλειας επιχειρήματα που ξεπερνούν το πλαίσιο το οποίο συζητούμε. Δηλαδή το πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, τα διαθωτικά ταμεία, τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνολικά. Αυτό ξεπερνά τα στενά πλαίσια στα οποία έχουμε τεθεί σήμερα. Όμως όπως προανέφερα Όλες οι αναλύσεις που κάνουμε είναι δημοσιευμένες, είναι δημόσιες, έχουν δημοσιοποιηθεί και μπορούν να ε, είναι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο πολλοί από εσά προανέφεραν είναι το θέμα της γραφειοκρατίας και η σύνδεση αυτού του ε, στοιχείου με το πρασίνισμα. Γι' αυτό επιλέξαμε όμως τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα μέτρα που επιλέξαμε, διότι είναι τα μόνα μέτρα τα οποία εντοπίσαμε που μπορούν να επιτευχθούν με ένα ελάχιστο ποσοστό επιπρόσθετου ελέγχου ή γραφειοκρατικού διοικητικού ε, βάρους ε, ως δαπάνη. Όλα αυτά θα πρέπει να, να πούμε ότι από πλευράς ε, του συστήματος είναι διαθέσιμα. Και στρέφομαι στο θέμα του κυρίου Λάιονς και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ε, εξαιρέσαμε το green cover, το, την πράσινη επιφάνεια ή επικράτεια. Διότι πώς μπορεί κανείς να ε, εντοπίσει ή να ταυτοποιήσει αν υπάρχει αυτή η ε, πράσινη έκταση. Οι διαφορές είναι πολύ βόρειων και νότιων χωρών και αυτό θα απαιτούσε επιπρόσθετους ελέγχους. Παρότι αυτό είναι ένα μέσο ένα εργαλείο που όλες οι περιβαλλοντικές αναλύσεις αποφαίνονται γι' αυτό ότι είναι εξαιρετικά θετικό και σε σχέση με τις επιπτώσεις και όρους ε, περιβαλλοντικής ε, επίπτωσης. Τώρα, πώς ε, αξιολογήσαμε σε σχέση με το κόστος και όχι αυτό σε σχέση με φήμες του 5%. Αναλύσαμε εξειδικευμένα ένα μέτρο και βλέπουμε ποιο είναι το πρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος όσον αφορά τα μέτρα πρασινίσματος, ακόμα και ε, την πράσινη έκταση green cover. Από αυτό πρέπει να αφαιρεθούν ε, άλλες δαπάνες απλούστευσης. Έχουμε λιγότερους κανόνες όσον αφορά λιγότερους κανονισμούς και πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τον πρώτο πυλώνα. Θα υπάρχει μία αρχή για τις πληρωμές σε όλα τα κράτη-μέλη μεγάλη απλούστευση που γίνεται και για το εγχείρημα για τους μικρογεωργούς όπου 30% των εποφελούμενων είναι 3%, καλύπτουν μόνο 3% της έκτασης και έτσι δεν επιβάλλεται σε αυτούς να επιβαρυνθούν γραφειοκρατικά με αυτά που θα επιβαρυνθούν άλλοι γεωργοί. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία υιοθετήσαμε και προ, ε, λάβαμε και υπάρχουν και πολλές άλλες ε, μικρολεπτομέρειες που αφαιρούνται από το συνολικό κόστος. Είναι ένας τομέας που εξετάσαμε πολύ προσεκτικά. Ερώτηση τώρα, γιατί πρέπει και χρειάζεται να εισαχθεί ένα, μια διαστρωμάτωση υποχρεωτικών δεσμεύσεων δεσμευτικών μέτρων πρασινίσματος στον πρώτο πυλώνα. Όταν υπάρχει η πολλαπλή συμμόρφωση ήδη και όταν υπάρχουν ήδη πρόσθετα κίνητρα εθελούς, εθελοντικού χαρακτήρα ε, όσον αφορά το γεωργικό τομέα στο δεύτερο πυλώνα. Και εδώ υπάρχει μια θεμελιώδης μετάθεση στη λογική προσέγγιση των πραγμάτων από πλευρά μας. Αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση για να σας δείξουμε το γράφημα που δείχνει όχι μόνο την αύξηση σε σχέση με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων, πράγμα το οποίο συμβαίνει παγκόσμια όπως και στην Ευρώπη, αλλά και την πολύ μεγαλύτερη αύξηση ε, κόστου στα παραγωγικά, ε, ε, στην παραγωγή προϊόντων, στην παραγωγική διαδικασία. Αν είναι μόνο η οικονομική ε, αηφορία που μετράει, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και παραγωγικότητας. Και αυτό σημαίνει να ε, προσαρμοστούμε σε σχέση με την ε, ε, ένταση της καλλιέργειας. Και αν έχουμε από την άλλη πλευρά οικονομική και περιβαλλοντική αηφορία που απαιτείται, πρέπει να υιοθετήσουμε και να εισαγάγουμε ένα τέτοιο συνδυασμό κινήτρων και περιορισμών, όρων και προϋποθέσεων που θα κινητοποιήσει τους γεωργούς να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι θα πρέπει να αντισταθμιστούν τα ωφέλη έναντι της επιβάρησης. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο κάναμε. Ίσως δεν το κάναμε με τον ιδανικό καλύτερο τρόπο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε προτάσεις για βελτιώσεις. Αλλά αξιολογήσαμε με, τις, με τον καλύτερο τρόπο και σε λεπτομέρεια τον κόστος το οποίο θα συνεπαγόταν αυτό, αυτές οι προτάσεις που θα συνεπαγόντουσαν και είναι σαφές από την ανάλυση ότι το δυναμικό, το ενδυνάμει ε, περιβαλλοντικό όφελος ε, που έχει ε, κατ' υπολογιστή και δεν ε, έχει υπολογιστή επιβάρυνση όσον αφορά την επιβάρυνση των γεωργών. Γι' αυτό κυκλοφορούν κάποιες φήμες σχετικά. Και γι' αυτό επειδή πολλά, όσα αφορά, πολλά από όσα αφορούν το κόστος δεν έχουν σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές της αγοράς και των εξελίξεων στη γεωργία, αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί εξωγενείς παράγοντες εκτός γεωργίας που διαμορφώνουν τις τιμές για παράδειγμα και των τροφίμων. Μπορεί να δείτε, μπορείτε να δείτε την τιμή του πετρελαίου και αυτό πάλι επηρεάζει τι γίνεται σε σχέση και με την μεθανόλη και άσχετα από ε, εκείνα τα οποία ε, εμείς είχαμε ε, ως θεμέλια για τους υπολογισμούς πριν από μερικά χρόνια. Και τώρα, βλέποντας το συσχετισμό μεταξύ των μέτρων πρώτου πυλώνα και δεύτερου πυλώνα, γενικότερα και τα, τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Αυτό που κάνει το πρασίνισμα είναι υποστηρίζει περιβαλλοντική υιοθεσία μέτρων παν, πανευρωπαϊκά στο, στο 50% τουλάχιστον των επιφανειών και βρίσκεται η δυνατότητα στοχοθετημένων μέτρων στο δεύτερο πυλώνα. Υπάρχουν εκμεταλλεύσεις οι οποίες ε, θα ε, υποστούν τις συνέπειες. Τώρα, τα κράτη-μέλη για τον υπολογισμό του πρόσθετου κόστους ε, που θα επιβαρύνεται μια, μια εκμετάλλευση ή απώλειες, ε, αλλά και αυτό θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε ευρέως ότι θα υπάρχει σημαντική επίπτωση ή σημαντική μείωση. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι η σύγχυση που δημιουργείται για το τι είναι δύο παρατηρήσεις. Η μία αφορά τις ε, οικολογικά επικεντρωμένες περιοχές. Να είναι σαφές αυτό, δεν έχει καμιά σχέση με την αγρανάπαυση, το set aside. Θα είναι περιθωριακές ε, εκτάσεις εκείνες ε, που ε, δεν θα καλλιεργούνται και η επίπτωση στην παραγωγή και παραγωγικότητα θα είναι χαμηλή, θα είναι μικρή. Και 5% ή στο 10% που αρχίζει να έχει επίπτωση μια, ένα τέτοιο μέτρο, γι' αυτό επιλέξαμε το 7%. Γιατί το κάνουμε αυτό. Το κάνουμε για λόγους βιοπικιλότητας και το κάνουμε επειδή μας είπαν και ενημερωθήκαμε επανειλημμένα και από τους συναδέλφους μας στη Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον και από περιβαλλοντικές ομάδες ότι πρέπει να δημιουργήσουμε διαδρόμους βιοπικιλότητας. Αν δεν γίνει αυτό, σε σχέση με μονάδες που ε, οδηγούνται στην αγρανάπαυση ε, περιθωριακών ε, ας το εκτάσεων που μπορούν να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση για να υπάρξει εξισορρόπηση θα πρέπει να ε, δούμε το τι είναι αναγκαίο να γίνει. Θα υπάρξει κόστος, ε, ναι, αλλά θα μπορεί αυτό να αντισταθμιστεί από τις καλλιέργειες ε, με τη βιοπικιλότητα που θα εισαχθεί. Θα υπάρχει βραχυπρόθεσμα κόστος, θα είναι, είναι σαφές ότι θα υπάρχει, αλλά μακροπρόθεσμα θα υπάρξει όφελος, είναι και αυτό σαφές. Ελπίζουμε, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμα όφελος με αυτά τα μέτρα. Και εν τέλει σε σχέση με τις ποσοστώσεις για τη ζάχαρη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πιστεύω ότι είναι η κατάργηση ποσοστώσεων το μέτρο εκείνο που θα επιτρέψει η παραγωγικότητα να αυξηθεί και να εξεταστούν άλλες εναλλακτικές δυνατότητες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα υπέρ και τα κατά ενός συστήματος. Ένα σύστημα προκαθορισμένης παραγωγής ε, σε σχέση με τις, ε, ε τιμές ε, που είναι ευμετάβλητες δεν μπορεί να περιορίσει τον ευμετάβλητο χαρακτήρα της κειμενόμενες τιμές. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό του εισοδήματος για τους γεωργούς που εκ προημίου θα είναι γνωστό ποιο θα είναι και μετά να μπορέσουμε να λάβουμε τα μηνύματα από την αγορά, να λάβουν οι γεωργοί τα μηνύματα από την αγορά, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο. Πρέπει με πολύ πιο στοχοθετημένο, καλύτερο τρόπο να γίνεται αυτό α, α, σήμερα. Και γι' αυτό θα πρέπει η περιφερική ανακατανομή να προβλέπεται α, όσον αφορά τα κράτη-μέλη, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε άμεσα. Σε σχέση με την ερώτηση που θέσατε εσείς, σε σχέση με το, την κλίδα κατανομής του δεύτερου πυλώνα, Κάναμε πολλές αναλύσεις. Η απόφαση του πώς θα γίνουν ε, αυτά τα πράγματα, μια και δεν έχω περισσότερα στοιχεία να σας αναφέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα συγκεκριμένο. Ε, ίσως έχω ξεχάσει κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο σας. Ξέρετε πάντα που, θα, που μπορείτε να μας βρείτε. Είμαστε πάντα πρόθυμοι και ανοιχτοί να υποβάλουμε περαιτέρω διευκρινήσεις αν χρειαστεί για να απαντηθούν ερωτήματά σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Τάσο Χανιώτη και τους άλλους συναδέλφους της Γενικής ως Άγκρη. Ξεκινήσαμε να εμβαθύνουμε στο περιεχόμενο. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αν δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος ο οποίος επιθυμεί να πει κάτι. Σημείο 5 λοιπόν. Τροποποίηση τη Οδηγία 2003-96 του Συμβουλίου σχετικά με αναδιάθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κ. Σεριο Γκουτιέρης είναι εισηγητής για την ομοδότηση. Η πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας όσον αφορά την φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων εισάγει ένα νέο σύστημα ελάχιστων ποσοστών ε, φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων επί τη βάση δύο συνιστοσών. Ενεργειακό περιεχόμενο ε, και εκπομπή διοξιδίου του άνθρακο. Η νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπεριέχει διάφορε διατάξει που συνδέονται συγκεκριμένα με το γεωρικό τομέα. Και γι' αυτό η Επιτροπή μας θεώρησε σκόπιμο να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Δίνω το λόγο στον Σέργιο Γκουτιέρες, υπενθυμίζοντας ότι η προθεσμία η υποβολή τροπολογιών είναι 29 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Μεταξύ μας υπάρχει και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Κολεσάνκα, που θα μπορούσε ενδεχομένω να απαντήσει τυχόν ερωτήσεις. Σέργιο, έχεις το λόγο. Sí, muchas gracias. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί μου, το κόστος της ενέργειας ε, είναι όλο και περισσότερο ποσοστό του παγίου ε, κόστος, κόστους της ερωτικές ε, μας εκμεταλλεύσεις. Βεβαίως το κόστος αυτό ποικίλει από κράτος σε κράτος, αλλά κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται στο 30% των παγίων εξόδων η πρώτη τροποποίηση της οδηγίας που έχουμε ενώπιόν μας τι προτείνει. Ένα νέο προσανατολισμό από τη φορολόγηση ε, για ε, την ενέργεια ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και το λεγόμενο ενεργειακό μείγμα ευνοούνται ε, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή άλλες πηγές και όχι τα ορυκτά καύσιμα με διπλή περίπου φορολόγηση και από την ενεργειακή τους ε, ε, δυνατότητα αλλά και επειδή παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε αυτό θα σημάνει αύξηση του παγίου κόστους της λειτουργίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων όταν γνωρίζουμε ότι ε, η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα τους έχει πολύ χαμηλά ε, περιθώρια για τους λόγους που γνωρίζουμε και είπαμε επιστημική ασφάλεια, κατάσταση στις αγορές κτλ. Και επιπλέον αν περιοριστεί ακόμα περισσότερο ε, το περιθώριο κέρδους τους όταν τεθεί σε ισχύ την 1η Πρώτου του 2013 αυτή η οδηγία θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που φοβούνται ότι θα χάσουν και τις άμεσες ενισχύσεις από τον πρώτο πυλόν. Έχουν γνωμοδοτήσει και άλλες επιτροπές όπως είναι η Επιτροπή Βιομηχανίας που ζητάει να ε, απαλληφθούν αυτά τα άρθρα που αφορούν τη διπλή φορολόγηση. Αλλά επειδή υπάρχει κίνδυνος ε, αυτές οι τροπολογίες όχι μόνο στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο διάλογο που θα γίνει στη συνέχεια με το Συμβούλιο και την Επιτροπή μπορεί να αναβαγίσουν αυτό που εμείς προτείνουμε είναι ε, να πούμε ποια θα είναι τα φορολογικά κίνητρα και οι ελαφρύνσεις που πρέπει να δοθούν στη Γεωργία γιατί δεν έχει ε, άλλη ε, λύση, άλλη επιλογή από τη χρήση ορυκτών καυσίμων για τη γεωργική παραγωγή. Έχουμε λοιπόν συνοψίσει ότι θα πρέπει να υπάρχουν χαμηλοί συντελεστές μέχρι και μηδενικοί στο πετρέλαιο το γεωργικό αφορολόγητα καύσιμα. Αν και η σημερινή διατύπωση στην οδηγία είναι πολύ αμφίσιμη. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια ή ασφάλεια δικαίου καλύτερα για τους γεωργούς μας. Γιατί εδώ υπάρχει μια αιρεσιμότητα ε, στις φορολογικές ελαφρύσεις ή και στις φοροαπαλλαγές σε σχέση με την απόδοση την ενεργειακή των εκμεταλλεύσεών τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε ένα στοιχείο εδώ ευελιξίας στους νέους ε, όρους, να μην είναι μεμονωμένες και ατομικές οι απαιτήσει, αλλά να είναι τακμηριωμένες, γιατί σήμερα δεν ξέρουμε πού βασίζονται, ούτε τι εξυπηρετούν. Να είναι λοιπόν κάτι ενταγμένο σε μια κρατική στρατηγική που να έχει σχεδιαστεί σε συμφωνία με τον κλάδο και να εκτείνεται σε αρκετά έτη για να μην είναι δυσβάσταχτο και επιπλέον φορτίο αυτό για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δεύτερος στόχος που ορίζουμε εμείς. Αφού τα κάνουμε όλα αυτά, δηλαδή και την ευελιξία και τους στόχους και τις εξαιρέσεις, σε σχέση με τα γιγατζάουλ. Αυτή η οδηγία επιτρέπει ε, σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα να επιβάλλεται φόρος ε, σε σχέση με άλλη οδηγία, τη 2003 87, που αναφέρεται στη λεγόμενη διαρροή διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή, να φύγουν οι ε, εκμεταλλεύσεις που παράγουν του διοξείδιου του άνθρακα. Υπάρχει ένα φύλλο πορείας για το 2050 ε, και αναγνωρίζεται και, η οδηγία, ε, και στην οδηγία αυτή ότι και η γεωργία ε, είναι ένας κλάδος που παράγει διοξίδιο του άνθρακα και κινδυνεύει από τη διαρροή και θα πρέπει να αλλάξει αυτή η οδηγία 2003 κάθετος 87 για να συμπεριληφθεί και η γεωργία ως κλάδο από τη διαρροή άνθρακα για να υπάρχουν αντίστοιχες διατάξεις και μέτρα και στη φορολογία. Και επίσης, πέρα από το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της γεωργίας, θέλησαμε να υπολογίσουμε και τι γίνεται με τη βιομάζα εδώ. Βεβαίως, αυτό βελτιώνει τη φορολογική αντιμετώπιση της βιομάζας είναι ευνοϊκή, αλλά θα πρέπει καλύτερα να οριστεί η βιομάζα. Δηλαδή, να μην έχουμε ένα ορισμό πάρα πολύ στενό ε, της έννοιας αυτή στην οδηγία και να αφήνει απ' έξω διάφορα στοιχεία βιομάζας ε, που είναι στο στάδιο της έρευνας ακόμα και επίσης θα καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση του ΦΠΑ Ξέρω ότι αυτό δεν είναι αντικείμενο της παρούσης οδηγίας, αλλά θα θεωρούσαμε πάρα πολύ σκόπιμο να ε, υπάρξει αντιστοιχεία στους συντελεστές ΦΠΑ για τη βιομάζα. Γιατί μας λέγουν από τον κλάδο ότι σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει μια κυκλοφορία παραμεθόρια όταν διαφέρει ο φορολογικός ε, συντελεστής ε, ε, όταν έχει υψηλό ΦΠΑ μια χώρα, πολύ μεγάλο συντελεστή, πηγαίνουν στη γειτονική. Λοιπόν, ε, στην έκθεση αυτή επίσης θα πρέπει να ενταχθεί και ένα σύνολο τροπολογιών που υποβάλλουμε εμείς ως Κοινοβούλιο και επίσης όπως δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, το σχεδιασμό και όλα τα στάδια. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας στόχη τελικά. Είναι μια έκθεση από τη φύση της πάρα πολύ τεχνική, αλλά δική μας είναι γνωμοδότηση. Bene, grazie. Ευχαριστώ τον Σέργιο Κουτιέρες. Ζήτησε ένας να πάρει το λόγο, Herbert Dorfman. Σας ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος επειδή με τα περισσότερα πράγματα τα οποία ο συνάδελφος προανέφερε συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό απόλυτα. Και η συνάδελφός μας η κυρία Λούλινγκ είναι η συγγήτρια στην αρμόδια καθήλυνη επιτροπή, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, την Οικονομική Επιτροπή και σίγουρα έτσι ε, μπορεί κανείς ε, να έχει μια συνολική επισκόπηση της πρότασης μια και βλέπουμε ότι στο Συμβούλιο δεν ε, προωθούνται αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα εδώ και μόνο επαναλήψεις μπορούν να γίνουν στα όσα προαναφέρθηκαν. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα η κατάσταση φορολόγησης των γεωργών όσον αφορά τα καύσιμα ή όσον αφορά τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία να μην ε, αλλάξει, να μην τροποποιηθεί εκ βάθρων. Αν τα συνδέσουμε αυτά με τα θέματα που συζητήσαμε τις τελευταίες δύο ώρες θα είχαμε μια ε, μεγαλύτερες δαπάνες ή μεγαλύτερη ε, επιβάρυνση φορολογική και αυτό θα ήταν καταστροφικό, θα ήταν ολέθριο για τους γεωργούς και σε σχέση με ε, με το καθεστώς που υπάρχει σήμερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αντιστάθμιση υπέρ των γεωργών και λαμβάνοντας υπόψη τη βιομάζα και φοβούμε όμως ότι σε σχέση με αυτή την πρόταση δεν υπάρχει περιθώριο για αλλαγή της οδηγίας ε, για το ΦΠΑ, εδώ μπορούμε να έχουμε κάποιους, ε, ε ας το πω έτσι, ευκταίους στόχους, ε, επενέσιμους στόχους, όμως δεν είναι δυνατό να αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά η βιομάζα και το θέμα της βιομάζας είναι ένα σημαντικό και θα γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα στο μέλλον. Και θα έπρεπε εδώ να πούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα οδηγηθούμε σε επιπρόσθετη φορολόγηση της βιομάζας που τελικά αυτό θα απέβαινε ε, ε, ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη βιομάζα. Κατά τα άλλα υποστηρίζω αυτά τα οποία μόλις προαναφέρθηκαν από πλευρά του εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χέρμπερτ. Μάρτιν Όσλιγκερ. Και εγώ θα ήθελα μια ερώτηση να διατυπώσω επειδή αναφέρεται σε κάποια παράγραφο τη βιομάζα, καταρχήν η, η, οδηγεί, η υποστηρίζει, η χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του άνθρακα. Δεν είναι αυτό υποχρεωτικό σε σχέση με, την, με τον αραβόσιτο ε, όταν υπάρχει αποθήκευση υπάρχει και απελευθέρωση. Κάτι άλλο θα έπρεπε να πούμε και να μην παραμείνει αυτό αναλύωτο έτσι όπως ε, έχει αυτό το εδάφιο. Εκείνο που με εκπλήσει είναι ότι δεν αναφέρεται κάτι το οποίο πολλοί έχουν ε, ε, πει σε σχέση με το ΦΠΑ. Έχουμε όμως και τελείως διαφορετική υποστήριξη της γεωργίας όσον αφορά την φορολογία, φορολογία του ντίζελ ως καυσίμου για τη γεωργία. Εδώ το γεγονός είναι ότι έχουμε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις στις χώρες μας ούτως ή άλλως. Όμως μακροπρόθεσμα οι στόχοι της διαμόρφωσης ε, της ενεργειακής πολιτικής ακόμα και αν είναι επενέσιμοι δεν θα πρέπει αυτοί να τίθενται στο επίκεντρο της ε, πολιτικής μας για τη γεωργία θα πρέπει να περάσουμε στην προώθηση των μη ορυκτών καυσίμων και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω να απουσιάζει εδώ κάπως Ξέρω ότι εδώ γίνεται λόγος ε, για τη γεωργία και την υποστήριξη του χύψη υπέρ της, ε, ε, των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, όμως θα πρέπει συνολικά να ακολουθήσουμε την προσέγγιση υποστήριξης μη ορυκτών καυσίμων. Και αυτό είναι μια κατεύθυνση που στην γεωργία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και σε σχέση με την φορολόγηση, χαμηλή φορολόγηση ή μη φορολόγηση των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάρτιν. Δεν έχει ζητήσει άλλο το λόγο, οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στην εκπρόσωπο. Α, η κυρία Λούλινγκ. Μετά. Μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώ. Το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την κυρία Κολεσάνκα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχαμε πρόθεση να πάρουμε το λόγο, αλλά θα προβούμε σε κάποια γενικά σχόλια όσον αφορά τι προταθήσει τροπολογία. Ευχαριστώ για, την, ε, τι απόψει και την ομοδότηση. Το νέο κείμενο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρέει σε μεγάλο βαθμό από την αναγκαιότητα μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακο. Αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλλαγή όσον αφορά την ε, γεωργία. Παρ' όλα αυτά, ο γεωργικός τομέας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει χαμηλότερες ε, ε, χαμηλότερους εντελεστές για καύσιμα για κινητήρε. Αναφέρθηκε ο συγκεκριτή και στη διαρροή του άνθρακα και την οδηγία 87 του 2003. Από ό,τι γνωρίζουμε, σε αυτό το στάδιο, η Γενική Διεύθυνση Γεωργία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί μελέτη επί του θέματο και τα μέσα 2012 θα βγουν τα πορίσματα για ενδεχόμενου τομεί ή υποτομεί τη γεωργία που θα θεωρηθούν ότι κινδυνεύουν από τη διαρροή άνθρακα. Όσον αφορά τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, ένας από βασικούς λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρεί την οδηγία είναι για να προσαρμοστεί και να διορθωθεί η ανισότητα που υπάρχει με τα βιοκαύσιμα. Η εθανόλη φορολογείται με τον ίδιο συντοντεστή όπως το πετρέλαιο. Και στο μέλλον τα μελλοντικά κείμενα δεν θα ισχύουν για βιοκαύσιμα που είναι βιώσιμα σύμφωνα με την οδηγία. Λοιπόν, έχουμε ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης. Τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν τα, δικ, τα δικούς τους εθνικούς συντελεστές σε σχέση με τα ελάχιστα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο ΦΠΑ καθορίζεται από, τον 2000, από τη 2006-112 την οδηγία και εναρμόνιση των συντελεστών ΦΠΑ δεν μπορεί να αποτελέσει τμήμα της ε, παρούσης προτάσεως. Η πρόταση αναφέρεται στον ορισμό της βιομάζας σε ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άρθρο 2, ε, ε της Οδηγίας 28 του 2009. Δεν υπάρχει ανάγκη για ειδικούς κανόνες για βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Τα κριτήρια ε, βιωσιμότητας είναι αυτά που ισχύουν. Η πρόταση αφορά μόνο τη φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων και δεν επηρεάζει τους ορισμούς των κρατών μελών για την βιομάζα που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της φορολόγησης. Υπάρχει και άλλη τροπολογία, η επαριθμόν 7 δεν αναφέρθηκε από τον εισηγητή, αλλά ίσως για να είμαστε σαφείς πρέπει να πω κάτι. Σύμφωνα με το άρθρο 5, 2 και 3 της Οδηγίας 2008-118, η οδηγία για την ενεργειακή φορολόγηση δεν ισχύει για τις Καναρίους νήσους, διότι υπήρξε η πρόταση ότι η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στι Καναρίους νήσους να εξαιρείται από τον φόρο. Η οδηγία δεν ισχύει αυτά και ευχαριστώ. Καλώ ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούλινγκ και μετά στο Σέργιο αν θέλει να δώσει απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πράδρε. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η συγκήτρια στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή που είναι καθήλυνα αρμόδια και θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι απλώς καλοπισμός ενός υφισταμένου κειμένου. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σκέτη επανάσταση. Ανακλούει η πυρήμνα είναι σαν τον Κοπέρνικο. Και μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Πρέπει να σας πω ότι οι απόψεις εδώ διαφέρουν και δίστανται πάρα πολύ μεταξύ των επιτροπών, αλλά όχι μόνο των επιτροπών, αλλά και μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Ας πούμε στην οικονομική και νομισματική, η σοσιαλιστική ομάδα έχει σκιώδη εισηγητή που είναι υπέρ και θέλει ακόμα περισσότερο, ενώ άλλοι συνάδελφοι θα κάνουν τροπολογίες για να ζητήσουν απλούστατα απόρριψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της πρότασής της ενώ, με την παρούσα ε, μορφή. Επίσης σημείωσα ε, και τη θέση των κρατών μελών όλα με λίγες εξαιρέσεις ε, πλην τριών έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Και θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη μας και τις πολιτικές πραγματικότητες. Εγώ ως εισηγήτρια είμαι σε μια πάρα πολύ δινή θέση τώρα. Θα πρέπει να περιμένω τις διάφορες νομοδοτήσεις, αλλά πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοι <coughs> δεν έχουν ακόμα κατανοήσει ότι όχι απλώς αλλάζει η προσέγγιση σε σχέση με τα ισχύοντα, γιατί μιλούν για ενιαίο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για τις εκπομπές οξυδίου του άνθρακα. Γίνεται λόγο για 20 ευρώ, οι πράσινοι συνάδελφοι το έχουν πάει ήδη στα 30 με ένα ελάχιστο συντελεστή φορολόγησης της ενέργειας που να επιβάλλεται σε κάθε ενεργειακό προϊόν. Εγώ κατά βάθο, ξέρετε, είμαι υπέρ αυτή τη προσέγγισης της ε, διότι θεωρώ ότι όταν φορολογούμε την ενέργεια με διπλό τρόπο και ως προς το διοξείδιο του άνθρακα και προς το ενεργειακό δυναμικό ε, είναι πιο λογικό σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση. Αλλά εκτός από την προσέγγιση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει και μια αναλογικότητα μεταξύ των διαφόρων πηγών ενέργειας. Και εκεί ακριβώς ε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Παράδειγμα, συγκεκριμένο, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υπάρχουν περισσότεροι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί του πετρελαίου σε σχέση με τη βενζίνη. Αυτή η αναλογικότητα θα πρέπει να διατηρηθεί. Δηλαδή, όχι μόνο στον ελάχιστο συντελεστή, αλλά και επειδή τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν πολύ ψηλότερους συντελεστές σε σχέση με τον ελάχιστο. Άρα θα κρυβίνει η ενέργεια και με τρόπο πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη Γερμανία 31 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου στη δίζελ. Βεβαίως θα υπάρξει και μεταβατική περίοδος, δεν λέω, αλλά αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα. πώς να το πω, Δεν έχει γίνει καμία μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη αντικτύπου στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον πληθωρισμό, διότι αυτό θα ε, επηρεάσει το σύνολο του κλάδου των μεταφορών. Αν αυξηθεί το κόστος του πετρελαίου, δίζελ. Και τα φορτηγά είναι πετρελοκίνητα. Τι θα τα κάνουμε. Εντάξει, μπορούμε να τα ε, ε, αλλάξουμε και να βάλουμε αέριο. Αλλά ε, τα τρακτέρ, οι γεωργικοί ελκυστήρες δεν είναι βενζινοκίνητοι, πετρέλαιο και είναι. Και θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τη γεωργία. Σε μεγάλο βαθμό βεβαίω απαλλάσσεται και εξαιρείται η Γεωργία, αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι σε άλλε επιτροπέ που θεωρούν ότι οι πάντε θα πρέπει να φορολογούνται και τι είναι αυτά τα πράγματα για τη Γεωργία γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αλλαγή της τιμής, η αύξηση του κόστους και ε, οι επιπτώσεις για το κλίμα. Στόχος ποιος είναι. Υπάρχει ένα στόχος για το 2020 για την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν υπολογίζουν καθόλου πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν τη γεωργική πολιτική, την αλληλευτική πολιτική, τη βιομηχανική πολιτική. Αφήστε δε και τον πληθωρισμό. Ήθελα να σας τα πω γιατί όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα, πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως από τη γνωμοδότησή σας. Και εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να αναμειγνύουμε ε, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης με το φόρο προστιθέμενης αξίας, μπορούμε να έχουμε ευσεβείς πόθους για εναρμόνιση του ΦΠΑ, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αν δεν έχετε ευσεβείς πόθους για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης, εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα. Ε, μία μόνο χώρα και είναι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, υπάρχει όπου το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη. Στις υπόλοιπες χώρες όχι. Θα πρέπει να το υπολογίσουμε, να δούμε πού θα μας βγάλει. Περιμένω και τις τροπολογίες. Ξέρετε, δεν είμαστε και στην απόφαση εδώ. Και χρειάζεται ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εκεί να είστε βέβαιοι ή τουλάχιστον θα πρέπει να ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη κατανόηση και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις για τη γεωργία. Για να αποφύγουμε τις ανητικές συνέπειες. Ανητικότατες θα έλεγα αυτής της πρότασης. Και για τις μεταφορές και για τη γεωργία αλλά και για τη βιομηχανία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Σέρχιο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι, συνοψίζοντας. Θέλω. Mm. Απλά θέλω να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν. Και για να τονίσω ένα από τα πράγματα που είπε η κυρία Λούλινγκ, διότι αληθεύει ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και το βλέπουμε αυτό, όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ομάδων, όλων των πολιτικών ομάδων και σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές τους επιτροπές που έχουν διαφορετικές θέσεις μεταξύ τους, αυτό είναι μία έκθεση, μία οδηγία που αφορά και θίγει πολλά συμφέροντα. Και γι' αυτό αληθεύει και είναι σημαντικό η συζήτηση που κάναμε σήμερα, συμμεριζόμενη τις φιλοσοφικές αρχές ε, επί της ουσίας για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας με τη γνωστοποίηση ότι φτάσαμε στο μέγιστο επίπεδο εκπομπών ρήπων διοξιδίου του άνθρακα και μας είπε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συζητήσουμε το θέμα της φορολογίας ενεργειακών φορέων στο ευρύτερο πλαίσιο. Και είναι σημαντικό να δούμε αυτό και ως ευθύνη μεταξύ της Επιτροπής Γεωργίας. Πρώτα, να προασπίσουμε τα συμφέροντα του τομέα, των γεωργών δηλαδή, της Γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη μια κοινή φιλοσοφία και κοινέ αρχές σε σχέση με την οδηγία αυτή για έναν απλό λόγο. Διότι η Γεωργία αφεαυτής ε, όντας θετική για τον έλεγχο όσον αφορά τις ε, εκπομπές ε, ρήπων και την καταπολέμηση των εκπομπών ρήπων με βάση τον τόνο, ανατόνο εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης όμως είναι ένας τομέας ο οποίος ε, πρέπει να συνεξεταστεί σε σχέση με αυτό το θέμα. Γι' αυτό η στρατηγική αυτής της έκθεσης είναι να προσπίσει τα δικά μας συμφέροντα των γεωργών. Πρώτον, επειδή είναι καλό για την αηφορία και τη βιωσιμότητα των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για την αηφορία, την ε, αηφορία των καλλιεργειών που πρέπει να συνεισφέρει και να είναι υπέρ των στόχων, της επίτευξης των στόχων αυτής της οδηγίας. Για το ε, ΦΠΑ πρέπει να πούμε ότι είναι μια σύσταση αυτό το οποίο ζητούμε και θέτουμε στην έκθεση. Δεν ζητούμε τροποποίηση που είναι θέμα άλλης οδηγίας. Θεωρούμε ότι η βιομάζα έχει επιπτώσεις και έχει μέλλον ως προοπτική και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια σύσταση από πλευράς της Επιτροπής μας να έχει επαρκή αντιμετώπιση παρόμοια αντιμετώπιση για να είναι αηφόρος ε, η βιομάζα στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Αυτό το οποίο προαναφέρθηκε αληθεύει μεν, αλλά εκείνο το οποίο μας ενέπνα είναι η φιλοσοφία της ε, οδηγίας. Αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή η οδηγία είναι να υπάρξει αντιστάθμιση σε σχέση με το πραγματικό κόστος σε σχέση με τις ε, δαπάνες για, την, ε, για τα καύσιμα. Ευχαριστώ όσον αφορά την υποστήριξη και από τη Γραμματεία και όσους συνεργάστηκαν από τη Σοσιαλιστική Ομάδα και προσβλέπω στις τροπολογίες και προτάσεις σας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την, οδηγία, την ε, έκθεση. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν στο Συμβούλιο για να προαχθεί, να προχωρήσει αυτό το θέμα, ευθύνη μας είναι να, ε, να προνοήσουμε ώστε να προχωρήσουν τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα όσο καλύτερα μπορούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σέρχιο ευχαριστώ όλους σας. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών για την έκθεση Γκουτιέρες είναι 29 Νοεμβρίου στις 12. Και τώρα πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού ΕΕΚ αριθμός 617-2009 του Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστοσης για τις αγωγές βοήου κρέατος υψηλής ποιότητας. Η συγγητής για την γνωμοδότηση είναι ο George Lyon. Περνάμε λοιπόν σε αυτό το σημαντικό θέμα. Συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Σε επαφέ ήρθαμε εκεί με τι Αμερικανικέ Αρχές. Ο εισηγητή είναι ο George Lyon. Υποστηρίζει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κανονισμό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί μια συμφωνία που προβλέπει δύο φάσει, σύμφωνα με τι οποίε η και ο Καναδά μειώνουν σταδιακά το επίπεδο των ε, και Ρώσων που επιβάλλονται στα προϊόντα της Ένωσης, ενώ η Ένωση αυξάνει σταδιακά την δρασμολογική της ποσόστοση όσον αφορά τα κρέατα υψηλής ποιότητας ανεφορμονών. Η και ο Καναδάς ήδη συμφώνησαν για πλήρη αναστολή όλων των κυρώσεων κατά της Ένωσης από τον Μάιο του 2011 ανοίγοντα στον δρόμο προς τα χεία εφαρμογή της δεύτερης φάση της συμφωνίας. Θα συμφωνείτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον George Lyon αν θέλει να μας ενημερώσει επί του θέματος. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ο κ. Κοτούρνη και άλλοι της Γενικής Διευθύνσεως ε, Γεωργίας και συνάδελφοι βεβαίως που μπορούν να πάρουν το λόγο αν επιθυμούν. Λοιπόν, θέλεις να πεις εισαγωγικά κάποια πράγματα, Τζορτ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την εισαγωγή. Καλύψατε τα περισσότερα σημεία που θα έπρεπε να αναφερθούν. Αξίζει τον κόπο να πούμε ότι διαπραγματεύτηκε η κάθε άστον αυτή τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να προσπαθήσει να διευθετήσει ε, τη διαφορά όσον αφορά τις ορμόνες του βοηού κρέατος που κράτησε πολλά χρόνια. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι η απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θεωρήθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες του ΠΟΕ και ότι δεν περάσαμε τα δικά μας επιχειρήματα στο πάνελ, στον που Επί μακρόν κράτησε αυτή η διαφορά και αυτή η συμφωνία προσπαθεί να επιλύσει άπαξ διαπαντός το θέμα. Όπως και ο φίλος μου ο Δεκάστρο ανέφερε, το πρώτο μέρος συμφωνίας ήταν 20.000 τόνοι αύξηση όσον αφορά την ποσόστοση για βόλιο κρέας εξαγωγές αμερικανικού κρέατος προς υψηλή ποιότητα προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και 68% των κυρώσεων είχε αφαιρέσει η Αμερική, η ΕΠΑ, εν μεταξύ αυτό το δεύτερο τμήμα αυξάνεται κατά 25.000 τόνους παραπάνω ακόμα ε, η εξαγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας από τη ΣΥΠΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν άρει όλες τις ε, κυρώσεις οπότε έχουν προχωρήσει κάπως περισσότερο όσον αφορά τη συμφωνία, την εφαρμογή της συμφωνίας οι Αμερικανοί το ερώτημα πώς να αντιμετωπίσουμε είναι τελικά είναι καλή συμφωνία ή κακή αυτή. Διότι η Επιτροπή έχει δυνατότητα να πει ναι ή όχι όσον αφορά το θέμα αυτό. Βλέποντα το θέμα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό κέρδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εγγυάται το δικαίωμα να διατηρήσουμε την απαγόρευση όσον αφορά εισαγωγέ ε, κρέατος βοήου που έχει ε, υποστεί επεξεργασία ε, με ορμόνες. Αυτό δεν συζητείται δεν απειλείται να σωρευτούν και άλλες κυρώσεις πέρα από τις κυρώσεις που θα μπορούσαν να είχαν επιβληθεί. Απαλλασσόμεθα από όλες τις κυρώσεις και στο μέλλον και από μελλοντικές κυρώσεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξει τη συμφωνία η Επιτροπή. Κά... Μια άλλη συνιστόσα που έχει μπει στη συζήτηση και θα, θα αναφέρω ότι την έθιξαν συνάδελφοι ε, στην προηγούμενη συζήτηση που έλαβε χώρα και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι σημειώσαμε δεόντω αυτά που υπόθηκαν. Προσπαθήσαμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή απάντηση όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν. Δεν νομίζω ότι ήταν σωστό να συσχετίσουμε τα δύο θέματα. Ε, ήταν δύσκολο. Αυτό που κάναμε τελικά, όπως εξήγησα όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση, όταν οι εκπρόσωποι αυτής της Επιτροπής συναντήθηκαν με τον κύριο Βόλσακ που ήταν Υπουργός Γεωργίας, και τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Κέρκ, δόθηκε υπόσχεση στην Επιτροπή ότι οι προτάσεις για νέους κανόνες για το πυρετός της ίπα θα δημοσιευόταν και θα γινόταν διαβούλευση πριν το τέλος του έτους. Οπότε ο υποφαινόμενος και ο συνάδελφος του ΕΛΚ, ο εισηγητής της Σύντρα είναι εδώ. με υποστήριξε και στείλαμε από κοινού επιστολή και εγώ σαν εισηγητή τη Επιτροπή μα και ο εισηγητή τη ΣΥΝΤΑ στον Τόμ Βούλσακ και του ζητούσαμε να επιβεβαιώσει γραπτό ότι πράγματι θα δημοσιεύσουν το νέο νόμο, το νέο νομοσχέδιο για την ε, κεφαλοπάθεια εγκεφαλοπάθεια προς ψήφιση στι ΗΠΑ. Και με, τον αρμόδιο επίτροπο, με τον κύριο Ντάλι, θα μα επαφή και μα υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προωθούσε το θέμα και το ζητούσε από την Αμερικανική κυβέρνηση όταν πήγε. Μέχρι τώρα δεν πήραμε απάντηση στην επιστολή που στείλαμε. Καθιστούσαμε σαφέστατο στι Αμερικανικές αρχές και στον Υπουργό Γεωργίας, τον είπα, και του αρμοδίου του Υπουργείου Γεωργίας ότι θέλουμε θετική απάντηση στην επιστολή, ούτω ώστε οι πολιτικέ ανησυχίε που εκφράστηκαν από τα μέλη τη Επιτροπή θα έχουν διασκεδαστεί επαρκώ και θα δοθεί απάντηση στι ανησυχίε και η υπόσχεση που μας έδωσε τότε ήταν ότι θα τιμήσει τις υποσχέσεις που έδωσε. Ευχαριστώ τους Κιώδης για τη βοήθειά τους και τις προσπάθειες που κατέβαλαν στο σημαντικότητα αυτό το ζήτημα και τη βοήθεια που έδωσε ο Γκονταλίφ, η σε μένα και ελπίζω τελικά να γίνουν αποδεκτέ οι συστάσεις μου για την αποδοχή αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Τζορτζ, Σμιτ και Μαγκίνες οι δύο μιλητές. Ευχαριστώ. Όλοι νομίζω συντομία μπορούμε να τοποθετηθούμε σε σχέση με την προσέγγιση που υιοθέτησε ο εισηγητής ε, να ε, ε, δεν είμαστε γραφειοκρατικό σώμα χωρίς φωνή που εγκρίνει εν τυφλό και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν κάτι δεν είναι βατό, τότε πρέπει να το πούμε και να το αναφέρουμε και πρέπει να διατηρήσουμε τη συζήτηση ε, ζωντανή να έχουμε όταν θα υπάρξει απάντηση στην Ευρωπαϊκή, στη, από την Επιτροπή σε αυτό το θέμα να μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια και είναι απόλυτα σωστό. Πρέπει να σημειωθεί οπωσδήποτε πρόοδο επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαγκίνε και Λεμπρούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον George Lyons για τη δουλειά που έκανε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ότι δεν ήμουν παρούσα όταν αρχικά συζητήθηκε αυτό το θέμα και βλέπω και κατανοώ το πώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα. Θα ήθελα όμως να καταχωρηθεί για τα πρακτικά, να καταχωρηθούν κάποιες ανησυχίες που έχω για κάποια από αυτά τα τεχνικά θέματα και για κάποια από τα, κάποια από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται. Και αναφέρεται ότι το θέμα αυτό τώρα μπορεί να ε, διευθετήσει το ζήτημα αυτό με αυτή τη συμφωνία. Σε σχέση όμως ε, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου του 2008 πρέπει να δούμε ότι μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται απαγόρευση για την εισαγωγή κρέατος που έχει ε, τα ζώα έχουν τραφεί με ε, ορμόνες. Είναι σημαντικό να αναφέρω το ότι σε σχέση με τις κυρώσεις κάποια από τα θέματα θα έπρεπε να ε, εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Όχι σε σχέση με τα συμπεράσματα αλλά με τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Οι Ιρλανδικές, τα ε, Ιρλανδικά στοιχεία ε, διαφέρουν σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην, ως ε, αριθμητικό μέγεθος στην έκθεση. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Συζητάμε αυτό το θέμα των εισαγών κρέατος ε, από το εξωτερικό στην Ένωση για το θέμα της αναλογίας, αναλογικότητας. Αν δει κανείς την υψηλή αξία αυτού του κρέατος για το οποίο κάνουμε λόγο, το 0,3% που εισάγεται ή και που μπορεί να καταλήγει στο 7,5% στο τέλος τέλος με τους δικούς μου υπολογισμούς. Προς όφελος ε, της διαφάνειας και της καθαρότητας θα έπρεπε να εξετάσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και θα έπρεπε να υπάρξει διασύνδεση σε σχέση με τα θέματα του αυθόδους πυρετού και της πογκόδους εγκεφαλίτιδας, εγκεφαλοπάθειας με, την, τα θέματα των εισαγόμενων αυτών κρεάτων. Καλό θα ήταν να υπάρξουν απαντήσεις. Ίσως θα έπρεπε να ξαναστείλετε μια επίστολη και ή να ζητήσετε να μας στείλουν με φάξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάποια απάντηση. Θα έπρεπε να είμαστε δίκαιοι και να επιμείνουμε να δοθεί αυτή η απάντηση και να μην αγοράσουμε γουρούνι στο σακί μην τα δεχτούμε όλα εν τυφλό. Και γι' αυτό θα έπρεπε να πούμε ότι θα αξιολογούσαμε αν γινόταν αυτό, θα το εκτιμούσαμε. Κατανοούμε βέβαια τα ευρύτερα πολιτικά ζητήματα, αλλά θέμα αυτής της Επιτροπής ε, δεν μπορεί να είναι να εγκρίνουμε χωρίς να έχουμε εξετάσει και συζητήσει πιο πριν. Ευχαριστώ. Λεμπρούν και Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κοιόδη συγγήτρια θα ήθελα να καλωσορίσω και να χαιρετήσω το συγητή για το έργο του καταναώ και του συναδέλφου, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας. Ακούστηκε αυτός ο όρος προηγουμένως, ακριβώς. Περί ευθύνης πρόκειται ο συμβιβασμό και η συμφωνία δεν είναι ποτέ συγκεκριμένη απάντηση σε ένα ιδεώδες. Να δούμε λοιπόν σήμερα με τη συμφωνία αυτή τι απαντήσεις έχουμε. Κατά την άποψή μου είναι ε, εντάξει, μέχρι και ικανοποιητικέ. Και είναι μια φάση των διαπραγματεύσεων που έχει οριστεί, έχει λήξει, έχει δρεωθεί και οι υφιστάμενες συμφωνίες ισχύουν. Νομίζω θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας και να θεωρήσουμε ότι είναι πρόοδος και μάλιστα σημαντική για αυτό το θέμα. Δεύτερον, στα πιάτα μας, τα δικά μας και των συμπολιτών μας, δεν θα έχουμε ποτέ κρέας με ορμόνες και αυτό είναι σημαντικό. Και κάτι, επειδή εδώ αυτή η ιστορία είναι πολλαπλή και έχει και τεχνικές πτυχές, Είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων που θέλουν ενδεχομένως περισσότερες διευκρινήσεις. Γιατί λέω ότι είναι πολλαπλή αυτή η προσπάθεια. Εκ των προτέρων, εγκρίνοντας αυτή τη συμφωνία, θα άρουμε ενδεχόμενες κυρώσεις ή φέρπουσες που θα μπορούσαν να μας επιβάλλουν. Τι σημαίνει αυτό. Είμαστε πλέον σε θέση και με όρους που βλέπουμε και κατανοούμε να προχωρήσουμε ε, και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις σε μια αγορά που είναι σημαντική. Και να καλύψουμε ένα χώρο ε, και μια αγορά που θέλει να αναπτυχθεί. Οι Ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι θα είναι λοιπόν σε καλύτερη θέση. Γνωρίζουμε την κατάσταση και θα πρέπει βεβαίως να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δώσουμε θετική γνώμη σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεμπρέν, Ελίζα Μπεθιέκερ και μετά Τζιμ Νίκολσον. Σε ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σε σχέση με τις παρεμβάσεις των συναδέλφων κατέστη σαφές ουσιαστικά και έχουμε θετικές πτυχές ε, από ό,τι αναφέρεται σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Εμείς ζητούσαμε πάντα να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές που θα ισχύουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας. Νομίζω αυτό καταφέραμε να γίνει και αποτελούν τμήμα των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων. Με ικανοποιούν τα όσα άκουσα. Ίσως θα μπορούσε να δώσει κάποιος μια απάντηση από τους συναδέλφους ε, που εξακολουθούν και ασχολούνται με αυτό το θέμα αυτής της συμφωνίας και είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα στοιχεία. Άκουσα ότι υπάρχουν λέει δυσκολίες με την παροχή αυτών των εισαγωμένων και μέχρι την Ευρώπη και τη Γερμανία, μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, λόγω του τρόπου με τον οποίο οι ποσοστώσεις αυτές αντιμετωπίζονται από πλευράς Ευρώπης. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε, όχι τώρα, εδώ και τώρα, αλλά στη Συμφωνία ΣΥΤΕΣ επαπειλούμενων ειδών, όταν κάνουμε τέτοιες συμφωνίες να υπάρχουν καλές λύσεις ε, ώστε να είναι θετικές ε, οι πτυχές αυτές για αμφότερες τις πλευρές. Ευχαριστώ Τζιμ Νίκολσον τώρα και μετά Κάπουλο Σάντος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι λακωνικότατος. Δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ τον εισηγητή ε, γιατί πολέμησε για μία έγκαιρη συμφωνία. Είναι καλή ώρα. Καλή στιγμή, αλλά συμφωνώ με εκείνου που αναφέρθηκαν στη διαφάνεια, στην ανοιχτή προσέγγιση και αυτό που να το προσέξουμε. Σε μεγάλο βαθμό ε, επιλύει τα προβλήματα που είχαμε επί μακρά περίοδο με τη ΣΥΠΑ. Καλό που λύνεται το θέμα τώρα και προχωράμε. Το τελευταίο που θα θέλαμε τώρα θα ήταν ε, να ακούγονται πολλά μεγαλόστομα λόγια από τη μια πλευρά και την άλλη. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε αυτή την εποχή. Συμφωνούμε λοιπόν με τον εισηγητή και να το στηρίξουμε στο Κοινοβούλιο. Επίζουμε και ο εισηγητής να πάρει την απάντηση περιμένει από την άλλη πλευρά. Και να δουν οι Αμερικανοί ότι και από εδώ υπάρχει θετική ανταπόκριση στην συμφωνία. Ευχαριστώ Τζιμ. Λουίς το γεγονό ότι είναι κανεί τελευταίο στο να παρεμβαίνει έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Ουσιαστικά όλα έχουν αναφερθεί. Θα ήθελα μόνο να πω στον συνάδελφο Τζορτζ ότι η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει απόλυτα την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Δεν ξέρω αν από πλευρά ε, Κοτούρνη θέλουν να δώσουν κάποιε λεπτομέρειε. Ο Δ. Κοτούρνη από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια και μετά να δώσω κάποιε απαντήσει στα τεθέντα ερωτήματα. Αυτά που ακούστηκαν στη συζήτηση. Τα δύο σχόλια πρώτα. Το πώ σημαντική είναι η συμφωνία. Είναι σημαντική διότι όπω αναφέρθηκε διατηρείται η απαγόρευσή μα όσον αφορά το βόλιο κρέα με ορμόνες. Σημαντικότατο αποτέλεσμα των συζητήσεων και των μακρών διαπραγματεύσεων με τι ΗΠΑ. Πάρα πολύ σημαντικό υπόθηκε θα το υπογραμμίσω εκ νέου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να διατηρηθεί αυτή η απαγόρευση. Δεύτερον, επιτρέπει η συμφωνία αυτή να βρούμε μία διέξοδο, να βρούμε μια τελική με τελικη ρυθμιση της διένεξης με τη ΣΥΠΑ. Δεν φτάσαμε ακόμα. Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί αυτό στην τρίτη φάση. Αυτό που σας ζητούμε να εγκρίνετε είναι να κινηθούμε προς τη δεύτερη φάση αναφέρθηκε, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω εκ νέου, ότι οι έχουν άρει τις κυρώσεις 13 μήνες πριν από το πρόγραμμα, από ό,τι προβλεπόταν. Θα έπρεπε 1η ε, Αυγούστου του 2012 να άρουν τις κυρώσεις. Το έκαναν πριν από το φετινό καλοκαίρι. Αυτό για μας δείχνει καλή πίστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να εφαρμόσουν αυτή τη συμφωνία, καλή την πίστη. Οπότε θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τα αντίστοιχα και να κινηθούμε προς τη δεύτερη φάση και ελπίζουμε ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για τελική διευθέτηση στην τρίτη φάση της διένεξης. Δηλαδή όταν φτάσουμε εκεί που θα λήξει αυτή η διένεξη και βέβαια και οι δύο διατηρούμε τα δικαιώματά μας στα πλαίσια του ΠΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που διαφάνει σαφώς από το Μνημόνιο συνεργασία. Δεν είναι ότι απεμπολούμε τα δικαιώματα στον ΠΟΕ, θεωρήσαμε ότι αυτή η διευθέτηση, αυτή η ρύθμιση μας οδηγεί από, σε μία λύση της διαφοράς και σε θετικότερο περιβάλλον όσον αφορά τη σχέση με τις ΗΠΑ. Όσον αφορά τη σπογκώδη εγκεφαλοπάθεια, ήδη αναφέρθηκε ότι ασκήθηκαν πολιτικές πιέσεις επί τον ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Επίτροπο Ντάλι και από τον συναδελφό του. Ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας παρέχετε κι εσείς είναι διοργανική αυτή η προσπάθεια εναντί των ΗΠΑ. Ευχαριστώ για τι επιστολέ που εσεί, ε, Πρόεδρε, έχετε αποστείλει μαζί με τον Πρόεδρο τη Επιτροπή ΙΝΤΑ και τον εισηγητή προ τον ε, Υπουργό Μπίλσεκ. Πρέπει να σα πω ότι ε, αργά προχωράμε, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν στείλει στον αρμόδιο φορέα για την ψήφιση του προπολογισμού το μέτρο, το αρμόδιο το δικό του, θα χρειαστεί τρει μήνε. Μέχρι τέλο Ιανουαρίου περιμένουμε λοιπόν ότι το πρώτο βήμα θα έχει ολοκληρωθεί και είπα μετά θα δημοσιεύσουν το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει προθεσμία δύο μηνών, 60 ημερών, όπου εκεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρα μπορούν να σχολιάσουν. Μπορεί να παραταθεί η περίοδος ανάλογα με τα σχόλια που θα επιδοθούν. Αυτό που είναι σημαντικό σήμερα είναι να πούμε ότι υπήρξε μετακίνηση των ΗΠΑ τελικά έχει φτάσει στο, στην υπηρεσία διαχείρισης οικονομικής στο νομοσχέδιο κινούνται τα πράγματα χάρη στην υποστήριξη και την πίεση που έχετε ασκήσει κι εσείς επί τον ΙΠΑ. Δεν γνωρίζω τα προβλήματα παράδεση που ανέφερε η κυρία Γέγκελ. Με τα χαράς όμως να το εξετάσω αυτό διμερώς μαζί σας ή αν θέλετε σε οποιοδήποτε άλλο βήμα και πλαίσιο που επιθυμείτε. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοτούρνη. Βίσταρ Χορόελ έχει το λόγο που είναι συγγήτρια για την γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ειλικρινά ομολογώ ότι είμαι παλιά καραβάνα εδώ στο Κοινοβούλιο και σπάνια έχω δει τόσο καλή συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Τζος Λάιον, εγώ δεν θα μπορούσα να γράψω καλύτερη γνωμοδότηση στη θέση του. Ε, συμφωνούμε πάρα πολύ, πράγμα που δεν είναι πάντα αυτονόητο. Είπατε τίποτα κύριε Πρόεδρε, όχι. Ε, χάρη Πρόεδρο αυτά. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο αυτό πάντα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Παρόλο που δεν σας γνωρίζω ε, αρκετά. Λοιπόν, 16 χρόνια διαρκεί αυτή η διαμάχη, καιρός να τελειώνει. Δύο-τρία σχόλια. Πρώτον, οι υπολογισμοί. Αν είναι 0,36%, 7%, αν ρωτήσετε δύο-τρεις άλλους εμπειρογνώμονες θα σας πούνε και άλλα στοιχεία. Και είναι και ο τρόπος υπολογισμού ε, σχετικός με την παρατήρηση, με το πώς το βλέπει καθένας. Εν πάση περιπτώσει δεν ε, αλλάζει σημαντικά η ε, κατάσταση με τα αριθμητικά στοιχεία. Ένα αυτό. Δεύτερο, σε σχέση με τη σκουπογκώδη εγκεφαλοπάθεια των βοηδών, στην αρχή είχαμε θεωρήσει ότι η αμερικανική αγορά θα μπορούσε ταυτόχρονα να ανοίξει και για τα δικά μας προϊόντα, αλλά τελικά δεν ε, πέρασε αυτό. Καλύτερα ε, να γίνονται ένα-ένα τα βήματα. Και σήμερα το μεσημέρι ε, μίλησα με εκπρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση της επόμενης συνεδρίασης ΤΕΚ το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου προφανές και αυτονόητο. Αυτό που έκαναν εκ των προτέρων και αποφάσισαν ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα χαιρόμουν αν ε, μπορούσαμε ε, γίνεται και ομόφωνα να αποφασίσουμε για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ και πάλι για την καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Μάριο, ε, κύριε Μαγκίνες, το λόγο. Ευχαριστώ που επιτρέψτε μου να διευκρινίσω με την εισηγήτρια κάποια στοιχεία, ίσως να μην χρησιμοποίησα σωστά τα στοιχεία. 0,36% της αγοράς βοήου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ανέφερα 7,5% ε, του, του, του κρέατος υψηλής ποιότητας. Αυτό και δεν αλλάζει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Μάριο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Δίνω το λόγο τον τελικό στον George Lyon. Για να συνοψίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη για τις απόψεις τους. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Ευχαριστώ τον κύριο Σμίθ για τα σχόλιά του. και είναι ενδεδειγμένο, είναι σωστό που συζητεί το θέμα τη πονκόδου εγκεφαλοπάθεια. Ναι, η απαγόρευση θα μπορούσε να παραμείνει, αλλά η, διαφορά με απειλή φερετέρω κυρώσεων ε, ε, ε, δεν θα επιλύει Η διαφορά είναι το θέμα. Η απαγόρευση α μείνει. Το 7,4% είναι σωστό το μερίδιο αυτό τη αγορά κρέατο ποιότητα. Σωστά το αναφέρετε. Εκτιμούμε ποιο είναι το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κρέατος ποιότητας. Τώρα τα στοιχεία όσον αφορά τα ωφέλη άρσης των ε, κυρώσεων, τα στοιχεία που αναφέρεται είναι οι τιμέ όταν πρωτοσύχθησαν οι κυρώσεις. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησαμε είναι οι τρέχουσες εκτιμήσεις των ωφελών για τα κάτι μέλη από την άρση των κυρώσεων σε σημερινές τιμές. Είναι διαφορετικά στοιχεία. Παρήγαγε επικαιροποιημένα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει όσο φανά την καθαρή αξία σε σημερινές τιμές των κυρώσεων. Και όχι την εποχή που επιβλήθησαν αρχικά οι κυρώσεις. Και αυτό το αναγνωρίζω και το λαμβάνω υπόψη. Ναι, να στείλω και άλλη επιστολή με τα χαράς. Από ό,τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει πρόοδος. Τουλάχιστον όταν πήγε στην αρμόδια υπηρεσία ε, την υπεύθυνη για τον προπολογισμό είναι δημόσιο στον ανοιχτό τομέα. Θα θέλαμε ο Επίτροπο Βόρσεκ να μα στείλει μια επιστολή και να μα πει ότι πράγματι συνέβη αυτό που είπατε και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει και με να του στείλουμε οτιδήποτε θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ε, τους ε, κάνει να τρέξουν εκεί. Συγγνώμη την ορολογία που χρησιμοποίησα. Να τους ρίξουμε νεύτη. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω ε, η Έσπεθ Γέγκελ αναφέρθηκε στο πώς λειτουργεί η διαχείριση των ποσοστών από πλευρά ΗΠΑ και Καναδά. Πώς λειτουργεί το σύστημα. 20% πρημοδότηση δίνεται στην τιμή απόκτηση αυτών των δικαιωμάτων βάσει του πώ εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσώστοση. Αντί ο δασμό να είναι 0 μέχρι 200%, η τιμή πληρώνει 20%. Από 0 μέχρι 20, αυτή πληρώνει 20% παραπάνω. τέλο πάντων, το συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε πώ εφαρμόζουν αυτή τι ποσοστώσει. Και ευχαριστώ του συναδέλφου για την έξοχη συνεργασία. Δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα για να το προωθήσουμε, αλλά ελπίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και επ' αυτού και επί της πογκόδους εγκεφαλοπαθίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζόρτζ, ευχαριστώ όλους. Πάμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για τη σημερινή συνεδρίαση. Πάμε λοιπόν στον εμβολιασμό κατά του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων. Εισηγητής ο Γιάννους Βοητσεβόσκη, ο Αντιπρόεδρος. Θα ήθελα να επενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι το Κοινοβούλιο θέτησε τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση από αυτού του θέματος τον Απρίλιο, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο λόγω μεγάλων διαφορών όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχειών. Πρόσφατα, οι διαπραγματεύσει οριζόντιου χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά το θέμα των πινάκων αντιστοιχία ε, κατέληξαν σε κάποια συνεννόηση και επιτευχθεί συμφωνία. Μετά από τη συμφωνία, το Συμβούλιο πρότεινε σε μια επιστολή στι 27 Οκτωβρίου που πέρασε ταχεία συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση του θέματος. Το κείμενο που πρότεινε το Συμβούλιο σας απεστάλει, σας έχει διανεμηθεί, οπότε δίνω λόγο, το λόγο στον κύριο Βουτσεβόσκι ε, για να ε, μας πει αν υπάρχουν κάποια καινούρια στοιχεία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα αυτό δεν μας απασχολεί για πρώτη φορά. Όπως θύμισε ο Πρόεδρος, τον Απρίλιο σε μια ταχεία διαδικασία εγκρίναμε αλλαγέ στην οδηγία ε, και τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο εύκολα και πιο καινούρια εμβόλια ε, κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που είναι μια πολύ σοβαρή ασθένεια. Και σύμφωνα με όλα τα μηνύματα και τα σημεία που είχαμε, θεωρήσαμε ότι θα αρχίσει ο εμβολιασμό ήδη από το 2011. Αλλά συγκρουστήκαμε με το Συμβούλιο, όχι η δική μας Επιτροπή, αλλά η νομική υπηρεσία ε, του Κοινοβουλίου με τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου για τους πίνακες ε, αντιστοιχίας. Για την παρακολούθηση ε, της υλοποίησης, της τροποποίησης της οδηγίας. Προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι κακή ιδέα των πινάκων αντιστοιχία, Νομίζω ότι αυξάνει όντως την, ε, ε, τη διαφάνεια του νομικού καθεστώτος που επικρατεί. Ωστόσο το Συμβούλιο ήταν ε, κάθετα αντίθετο και η οδηγία αυτή δεν τέθησε σε ισχύ την ημερομηνία που είχε προβλεφθεί αρχικά. Οπότε η θέση μας τώρα είναι να εγκαταλείψουμε τους πίνακες αντιστοιχίας, γιατί δεν είναι αυτό κρίσιμο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συντομότερο να εγκριθεί η οδηγία για να μην χάσουμε τη νέα περίοδο εμβολιασμών. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Εργαστήκαμε πάρα πολύ γρήγορα για να προετοιμάσουμε όλες τις απαραίτητες προτάσεις και πάλι είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Βοητσοκόφσκι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν να πούν τίποτα. Τίποτα. Όχι, λοιπόν. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, πάμε το ταχύτερο δυνατόν στην σύναψη συμφωνήσεων αφορά τη δεύτερη ανάγνωση και θα θέσουμε τη λέξη τέλος όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά του καταλογικού πυρετού του προβάτου. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να μιλήσουν, εγώ θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μα σήμερα. Τη Επιτροπή να υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί στι 9 θα κάνουν πρώτα τη συνεδρίαση των συντονιστών και από τι 9.45 θα ξαναρχίσουν τι εργασίε τη Επιτροπή με το σημείο 10 τη ημερήσια διάταξη.